Αγαπητές φίλες και φίλοι, παρακαλώ ε, να πάρει ο καθένας τη θέση του για να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα πραγματικά να, να ευχαριστήσω και το, το Policy Department και την ε, γραμματεία της, ε, ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διοργάνωση αυτής της συζήτησης για δεν το γνωρίζετε, αυτή η συζήτηση έχει το χαρακτήρα της διαβούλευσης μέσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και την ευρύτερη διαβούλευση με ε, τους, τα υπόλοιπα όργανα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ε, θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους φορέων. Είμαι ο Κρήτο Αναστέρης, είμαι ο της έκθεσης ε, για τα δάση και την προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή. Θα μιλήσω πολύ σύντομα πριν ε, ε, αρχίσουμε να περάσουμε στο πάνελ των ομιλητών και πραγματικά ακούσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν να μας πούνε. Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε είναι τα δάση. Και ο καθένας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, έχει μια μοναδική ιδιαίτερη προσωπική σχέση με τα δάση. Είναι στοιχείο της πολιτικής, πολιτικής κληρονομιάς του καθενός μας ξεχωριστά, είναι στοιχείο της ιστορίας μας του καθενός μας ξεχωριστά, είναι στοιχείο της οικονομίας μας του καθενός μας ξεχωριστά και είναι και ένα στοιχείο πολλές φορές της ε, καθημερινότητάς μας, ε, του χώρου στο οποίο βρισκόμαστε, της ταυτότητάς μας. Για όλους μας, για κάθε έναν Ευρωπαίο πολίτη, τα δάση είναι μοναδικά, σημαντικά και αναγκαία. Την ίδια στιγμή όμως, όταν μιλάμε για τα δάση, ο καθένας από εμάς αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό. Βρίσκονται, κάθε χώρα της Ευρώπης βρίσκεται σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, αν θέλετε. Βρισκόμαστε σε διαφορετικές περιοχές. Τα δάση μας έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δάση της ε, Νότιας Ευρώπης, της Μεσογείου, της Ανατολικής Ευρώπης, διαφορετικά τα δάση των Άλπαιων, διαφορετικά της ε, Κεντρικής Ευρώπης και πολύ διαφορετικά επίσης και τα δάση ε, στην βόρεια εποχή της Σκανδιναβίας, κοντά, πιο κοντά στους πόλους. Είναι διαφορετικά και αυτό σημαίνει ότι έχουν και διαφορετικές χρήσεις πολλές φορές, έχουν διαφορετική μορφή, διαφορετικές απειλές και ανάγκες. Όμως υπάρχει κάτι κοινό για όλα τα δάση. Αρκετά, αλλά ένα πάρα πολύ βασικό. Και είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συζήτηση, με την ευκαιρία της έκθεσής μας για την ε, προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή. Είναι μια κοινή απειλή. Η απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η απειλή αυτή ε, έχει και διαφορετικές διαστάσεις, που σημαίνει ότι σε κάθε βιοκλιματική ζώνη θα υπάρξουν διαφορετικές, ε, διαφορετικές είδη ε, απειλής, διαφορετικά, διαφορετικές απειλές και διαφορετικές ανάγκες προσαμωγής πολλές φορές, όμως έχει και κοινά. Ε, Κοινέ απειλέ φέρνει η κλιματική αλλαγή, όπως είναι βέβαια οι καινούργιες αρρώστιες των δασών που μεταφέρονται από μια χώρα στην άλλη, σε περιοχές που δεν υπήρχαν πρωτήτερα ε, και πάρα πάρα πολλά άλλα. Με όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα κοινό, τα δάση και το πόσο σημαντικά είναι αυτά για μας. Είμαστε σε διαφορετικέ περιοχέ, με διαφορετικέ ανάγκε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όμω έχουμε την κοινή ανάγκη να προσαρμοστούμε σε αυτή την απειλή. Και έχουμε και κοινέ απειλές που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Έχουμε οπότε ανάγκη τόσο πολύ, τόσο για ε, τη διατήρηση ε, δυνατοτήτων παρέμβασης σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά τις επιλογές μας για τα δάση και πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις κοινέ απειλές, όσο όμως και την ανάγκη για να χαράξουμε κοινέ κατευθύνσεις και να δούμε από κοινού πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν θέλω να μακρηγορήσω, είμαι εδώ πέρα για να ακούσω. Είμαστε στην διαδικασία προετοιμασίας της έκθεσης του Κοινοβουλίου για την ε, ε, προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή. Είναι, κρίσιμο, ε, είναι κρίσιμες η, η, συμμετοχή και η συμβολή σας σε αυτή τη συζήτηση. Ανυπομονώ πραγματικά να ακούσω το καθένα σας ξεχωριστά και τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους τη γνώμη για αυτό το θέμα, τι θα χρειαστεί να κάνουμε όσον αφορά την παρακολούθηση των δασών, ένα κύριο ζήτημα. Τι χρειάζεται να κάνουμε για την προστασία των δασών, για το θέμα των πυρκαγιών και τόσα άλλα κοινά ζητήματα. Και τι άλλα εργαλεία πολιτικής θα πρέπει να ετοιμάσουμε, να χαράξουμε ε, και να συναποφασίσουμε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρουσιάσω το πάνελ των ε, εκλεκτών ομιλητών. Στα δεξιά μου βρίσκεται ο κύριος Χάμελ, ε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, επικεφαλής ε, της, ε, του τμήματος της διεύθυνσης περιβάλλοντος που ασχολείται με τα δάση και με άλλα θέματα, αλλά είναι το τμήμα που, από την Περιβάλλοντος που ασχολείται και με τα δάση. Ε, επίσης μαζί μας είναι ο κύριος, ο κύριος Μάρκος, Μάρκος Λίντεν. Ε, ο κύριος Λίντεν έχει εκπροσωπεί την ομάδα την επιστημονική που ετοίμασε την έκθεση εκ μέρους της Διεύθυνσης ε, αγροτικών, αγροτικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισήγαγε, αν θέλετε, και αυτή την έννοια ε, έτσι πιο, πιο οργανωμένα την έννοια των πέντε βιοκλιματικών ζωνών. Και θα ακούσουμε με πολύ προσοχή αυτά που έχει να μας πει επίσης. Παρόν είναι επίση και ο κύριο Βίνκελ, ο οποίο θα συμμετέχει στη συζήτηση. Ο κύριο Βίνκελ εκπροσωπεί την ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, που ετοίμασε την έκθεση που ήταν ε, η βάση για την πράσινη ε, βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή. Ε, θα ακολουθήσει, θα υπάρξει ένα μικρό διάλυ, μια, μια μικρή ε, ευκαιρία για ερωτήσεις για 20 λεπτά και συνέχεια θα προχωρήσουμε στο δεύτερο πάνελ που θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ζακλή Μακλέιτ ε, που βρίσκεται επίσης στα δεξιά μου ε, η κυρία Μακλέιντ είναι η επικεφαλής, είναι η, ε, η διευθύντρια του European Environmental Agency της Ευρωπαϊκής Αρχής για το Περιβάλλον ε, με πάρα πολλή δουλειά και γνώση για τα θέματα της σημασίας των δασών για την δέσμευση των κλιματικών εκπομπών και την συμβολή των, των δασών της απειλές των δασών από τις αλλαγές χρήσης ε, αλλά και τη συμβολή του και τη σημασία του για την κλιματική αλλαγή. Όπως ε, επίσης ο κύριος ε, Μπερνάντε Καλεμπέρ, που βρίσκεται εδώ πέρα επίσης, εκπροσωπεί ένα πολύ σημαντικό κλάδο παραγωγικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την, της βιομηχανίας χαρτιού και είναι εδώ πέρα να μας παρουσιάσει την άποψη των παραγωγικών κλάδων για αυτή την απειλή και το τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Όπως επίσης η κυρία Βέλε Ντόσε από την, που ε, ε, θα εκπροσωπήσει κοινά με την παρουσίασή της την ε, Fern και την BirdLife, την ορνηθολογική, δύο οργανώσεις με πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και δράση στα θέματα των δασών και την προετοιμασία τους και την προστασία τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Δεν θα πάρω άλλο χρόνο, θα δώσω κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Χάμελ. Mr. Χάμελ, you have the floor. Thank you very much. Thank you. Ευχαριστώ. Καταρχάς, δηλώνω ότι ε, προπαρασκευάζοντας αυτό το κείμενο, η Κομισιόν ήθελε να ξεκινήσει μια συζήτηση για τις δυνατότητες που έχουμε να προστατεύσουμε τα δάση και να ενημερώσουμε το θέμα αυτό. Θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια συζήτηση κάθε παρέμβαση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα δάση με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμη η αρχή αυτή. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι να επιτεθούμε, να παραβιάσουμε την επικουρικότητα, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν τα κοινοτικά όργανα να βοηθήσουν ούτω ώστε να ενισχυθεί η προστασία των δασών μας λόγω των προκλήσεων που προκαλεί η, η κλιματική αλλαγή. Και τι ανάγκες ενημέρωσης υπάρχουν. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να υπάρξει επικοινωνία και η πράσινη βίβλος που ετοιμάσαμε πρέπει να αντιμετωπιστεί από αυτό το πρίσμα. Βάση μας είναι το σχέδιο δράσης για τα δάση, η στρατηγική μας για τα δάση και η λευκή βίβλος για την προσαρμογή. Αποτελούν το πλαίσιο. Αυτή η πράσινη βίβλος όμως, που νομίζω ότι είναι το πρώτο αρκετά σημαντικό κείμενο για τα δάση εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν το κείμενο στοχεύει στο να ξεκινήσει μια συζήτηση μέσω της οποίας και η Επιτροπή αλλά και άλλοι θα εγκρίνουν ιδέες και θα προχωρήσουν στη δράση τους. Αλλά θα μιλήσω αναλυτικότερα γι' αυτό. Το έγγραφο αυτό έχει υποβληθεί εδώ και 8-9 μήνες περιγράφει την κατάσταση, περιγράφει τη σημασία των δασών, τη λειτουργία τους, τις προκλήσεις και κάνει και μια επισκόπηση των δυνατοτήτων που έχουμε σε κοινωτικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και θέτει και μια σειρά ερωτήσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια ούτως ώστε να έχουμε υψηλή αποτελεσματικότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είμαστε τόσο σημαντικοί, μόνο 5% των δασών έχουμε. Άρα πρέπει να δούμε τη σφαιρική προσέγγιση και το κείμενο αυτό ασχολείται με την ε, συνολική, την ε, παγκόσμια προσέγγιση. Ποιες είναι οι λειτουργίες τώρα. Ως Επιτροπή θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε την κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική πλευρά της λειτουργίας των δασών, τους ώστε κάθε τομέας δραστηριότητας, κάθε συμφέρον που ασχολείται με τα δάση, να μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο, να μπορεί να λειτουργήσει, να μας πει αν εκπροσωπείται σωστά στο πλαίσιο που δημιουργούμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για λειτουργίες λοιπόν, των δασών, πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τις, ασχολούμεθα με τις οικονομικές λειτουργίες δηλαδή τις επιπτώσεις στην άμεση και έμεση απασχόληση και τον κύκλο εργασιών που προκύπτει, το ύψος του κύκλου εργασιών. Αυτές είναι σημαντικές λειτουργίες των δασών και οπωσδήποτε θα ε, φυγούν από την ε, κλιματική αλλαγή. Άλλη κοινωνικο-οικονομική λειτουργία των δασών είναι βεβαίως η προστασία για οικισμούς και για υποδομές, για παράδειγμα στη Γαλλία και στην Αυστρία, όπου έχει μεγάλη σημασία αυτή η λειτουργία των δασών. Από την αρχή λοιπόν εμένουμε στις κοινωνικο-οικονομικές πλευρές των δασών. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε σε ισορροπία με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα δάση προστατεύουν τα εδάφη. Τα δασικά εδάφη γενικά έχουν υψηλότερο, υψηλότερη περιεκτικότητα σε διοξίδιο του άνθρακα από τις γεωργικές γέες και είναι πιο σταθερά εδάφη. Έχουν ρόλο τα δάση στην ρύθμιση της παροχής του ύδατος. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν καθορίσει ορισμένες περιοχές όπου δίδεται πρωταρχική σημασία σε αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, και αναφέρατε στο κείμενο, η Γερμανία και η Ισπανία. Πρωταρχική σημασία έχουν ε, τα ευρωπαϊκά δάση για την βιοπικιλότητα. Έχουμε λοιπόν τη σχέση ανάμεσα στην βιοπικιλότητα, Natura 2000 στην Ευρώπη, με τα δάση. Τονίζουμε λοιπόν την περιβαλλοντική λειτουργία αυτή των δασών. Τέλος, τα δάση αποτελούν αποθήκες, αλλά και βέβαια και πηγές άνθρακα. Σημαντικό στοιχείο. Τα δάση μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο και σημαντική δυνατότητα, δώρο θα λέγαμε, για να αποθηκεύσουμε διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό όμως θα φυγεί από την κλιματική αλλαγή από την επέκταση της χρήσης της βιομάζας. Θα θυγεί. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την πρόκληση. Επίσης τα δάση παίζουν ρόλο στο περιφερειακό αλλά και τοπικό κλίμα. Το έχουμε τονίσει αυτό. Για παράδειγμα, τα δάση του Αμαζονίου παίζουν τεράστιο ρόλο στη ρύθμιση των βροχών δεν ξέρουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό το μέσο η Τζάκη να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς παίζουν τα δάση αυτό το ρόλο του στην Ευρώπη. Αυτό το ρόλο στην Ευρώπη. Όσο λοιπόν αναπτύσσεται περαιτέρω η δασική οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να δούμε ποια αντίμετρα πρέπει να έχουμε. Οι λειτουργίες λοιπόν αυτές πρέπει να εξεταστούν από πλευράς κλιματικής αλλαγής τι προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν οι λειτουργίες αυτές από την κλιματική αλλαγή, τι λειτουργία, τι κατάσταση θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε για την ανάπτυξη των δασών. Η πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι θα υπάρξουν ωφέλη σε περιοχές πιο βόρεια και σαφή, σαφή ζημίες ε, στις νοτιότερες περιοχές. Θα είναι δε πολύ ορατά τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής τα επόμενα 20-30 χρόνια. Και ήδη σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης είναι ήδη σαφή αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μιλάω τώρα για τις πυρκαγιές, μιλάω για την αποδάσωση, την αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθήκων, το θέμα των θυελών. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το θέμα των καταιγίδων. Ξέρουμε όμως ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής θα έχουμε όλο και περισσότερες καταστροφικές καταιγίδε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα προβλέψουμε, πού θα συμβαίνει, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις προστατεύοντας τα δάση μας. Και φυσικά και οι πυρκαγιές, οι δασικές πυρκαγιές. Κάνουμε τεράστια δουλειά και τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή τεράστιο όγκο δουλειά για τις ε, πυρκαγιές των δασών μαζί με πολλούς άλλους. Αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μας, κοστίζουν 1,5 δις ετησίως ευρώ. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα επιδεινωθεί το πρόβλημα αυτό των πυρκαγιών όσο αλλάζει η θερμοκρασία, οι συνθήκες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κατάσταση που είναι ήδη άσχημη. Ακόμη, στο κείμενό μας εξετάζει τα μέσα που έχουμε ως Ένωση. Έχουμε την επιτήρηση που έγινε μεταξύ 86-87 με 2006. Έχουμε την έρευνα που έχει γίνει, πολλές μελέτες Έχουμε την επιτήρηση των πυρκαγιών, ανάπτυξη της υπαίθρου. Προσπαθούμε να δώσουμε μια εικόνα στο πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι μπορούμε να επιτύχουμε. Με βάση, όπως είπα, ήδη από την αρχή, την επικουρικότητα. Να επανέλθω τώρα στις ερωτήσεις που έχουμε εδώ στο στο κατάλογο εδώ μπροστά μου. Ήδη με πολλές έχω ασχοληθεί. Υπάρχουν ε, πέντε ερωτήσεις που μερικές τις έχουμε, κάνει, ε, έχουμε χωρίσει και σε υποερωτήσεις, αλλά επειδή είμαστε διοικητικοί πάλι και θέλουμε να περιπλέκουμε τα πράγματα, το κάναμε αυτό. Πρώτον, το έγγραφο αυτό περιγράφει σωστά και ισορροπημένα τις λειτουργίες ε, των δασών. Οι ασχολούμενοι στον τομέα είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε σύντομα να δράσουμε. Είναι επαρκείς οι πολιτικές μας. Πώς να τις βελτιώσουμε αν δεν είναι. Η βιώσιμη διαχείριση των δασών πρέπει να ενημερωθεί ή είναι αποδεκτή όπως είναι. Μπορούμε να τη βελτιώσουμε από πλευρά κλιματική αλλαγής. Και ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση. Καλή, άσχημη. Πριν περάσω στις απαντήσεις, γιατί το κείμενο αυτό θα το παρουσιάσουμε στην μόνιμη Επιτροπή Δασών αύριο. Η Προεδρία, η Ισπανική Προεδρία ε, διατύπωσε τα συμπεράσματά της τον Ιούλιο. Περιμένουμε την ερχόμενη άνοιξη τα απορίσματα του Κοινοβουλίου και βεβαίως υπάρχουν και οι... αυτά τα κείμενα αλλά και οι απαντήσεις των εμπλεκομένων θα μας βοηθήσουν όλων των εμπλεκομένων φορέων θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω δουλειά μα. Αλλά δούμε τι απαντήσεις έχουμε. Ποιοι έχουν απαντήσει σε ερωτήσει μας. Λάβαμε 262 απαντήσεις συνολικά από τους, την, ε, τον κλάδο, από τις κυβερνήσεις, από μη κυβερνικές οργανώσεις, από τους ιδιοκτήτες και από εκλεγμένα σώματα και κοινοβούλια. Δεν είναι βέβαια στατιστική ανάλυση αυτή αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μέσω αυτής της διαβούλευσης, μέσω διαδικτύου, είχαμε αρκετές απαντήσεις από ενδιαφερόμενους υπεύθυνους φορείς. Εδώ βλέπουμε ποιοι δουλεύουν το καλοκαίρι. Γιατί αυτή η διαβούλευση ξεκίνησε αρχές του καλοκαιριού και τελείωσε τέλος καλοκαιριού. Τι περίεργο, οι Γάλλοι εργάζονται σκληρότερα από όλους το καλοκαίρι. Θα χαίρονται οι Γάλλοι συναδελφοί μου που τα ακούνε. Πολλές απαντήσεις από τη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία, Σουηδία. Βέβαια δεν μας εκπλήσει ότι έχουν πολλά δάση αυτές οι χώρες. Ενδιαφέρον ωστόσο ότι υπήρξαν απαντήσεις και από πολλές άλλες χώρες. Πού συμφωνούν λοιπόν, πού υπάρχει σύγκληση απόψεων. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη εναρμονισμένης ενημέρωσης για τα δάση. Ναι, είναι λίγες λέξεις, αλλά πίσω από αυτές τις λίγες λέξεις υπάρχουν 4-5 χιλιάδες κείμενα δυσπρόσιτα τα περισσότερα να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε την έρευνα για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στα δάση. Να διατηρήσουμε τον γονιδιακό πλούτο των δασών. Ενδιαφέρουσα άποψη. Να τονίσουμε σε ποιες περιοχές έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Στην ε, μεσογειακή ζώνη με τις πυρκαγιές. Και να συνεχίσει η κοινοτική ενίσχυση για την πραγματική ανάπτυξη πέθρου και για τα δάση. Εδώ λοιπόν συμφώνησαν γενικά οι συμμετέχοντες στην έρευνα και άμα διαβάσετε τα πορίσματα του Συμβουλίου είναι παρόμοια. Άρα συμφωνούν οι δύο αυτές πλευρές αλλά και για τις διαφορές συμφωνούν σε ποιους τομείς υπάρχουν αποκλήσεις απόψεων. Προφανής ο πρώτος τομέας. Αυτό το χάσμα ανάμεσα σε μια κοινοτική πολιτική που δεν την προτείνουμε φυσικά, είναι πράσινη βίβλος, και την επικουρικότητα. Επειδή είμαι υπεύθυνο και για τις γέες, Ξέρω και τον ορισμό αλλά και τι σημαίνει ο ορισμός. Το θέμα αν προστατεύονται τα δάση μέσω της διατήρησής τους στην φυσική τους κατάσταση ή μέσω της χρήσης. Βεβαίως και αυτό δεν μας εκπλήσει όταν ε, ε, απευθυνόμαστε σε όλους. Επίσης, πρέπει να εντείνουμε την εκμετάλλευση στην διαχείριση, να είναι έντονη η παρέμβαση ή να είμαστε ε, να αντιμετωπίζουμε τα δάση χωρίς να αποκλίνουμε από τη φυσική τους κατάσταση. Βεβαίως να χρηματοδοτείται η προσπάθεια αυτή, αλλά να μην υπάρχει νομοθεσία. Θα θυμάστε αυτά που έλεγαν οι άπικοι στην ε, Βόρεια Αμερική πριν από δύο αιώνες, ότι δυόμιση τώρα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση. Νομίζω ότι και εδώ θα μπορούσαμε εύκολα να διατυπώσουμε ένα ανάλογο σύνθημα. Και σε ποιο επίπεδο πρέπει να δρούμε. Είναι σε τοπικό, εθνικό, κοινοτικό, παγκόσμιο. Ποιο είναι το σωστό επίπεδο. Δεν υπάρχουν διαφορές. Αυτά λοιπόν μας λένε οι φορείς. Στο χώρο μας θα τα ε, παρουσιάσουμε όλα αυτά με πολλές λεπτομέρειες. Ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα. Πρώτα απ' όλα το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Θα υποβάλουμε έκθεση το 11 στο Συμβούλιο που να συνοψίζει όλα τα συμπεράσματα και κατόπιν και μετά ε, θα δείτε ότι λέμε ενδεχομένω ενδεχομένω σημαίνει δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε λοιπόν ε, τι θα προτείνουμε, τι δεν θα προτείνουμε. Ίσως κάτι για την ενημέρωση για τα δάση. Αν έτσι μας προτείνουν τα κράτη-μέλη, οι φορείς, το Κοινοβούλιο. Αν μας το προτείνουν θα το κάνουμε. Και αυτό θα προκαλέσει μια ε, νομοθετική πρόταση ε, κατόπιν. Θα δούμε. Η συμβολή λοιπόν της ε, συζήτησης που κάνουμε τώρα και του ψηφίσματος θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ιδέες μας το πρώτο εξάμηνο οκτάμινο του 11 γιατί στα πλαίσια αυτά πρέπει να αποφασίσουμε μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου για να ξεκινήσει η σοβαρή προσπάθεια με όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, παντού στην Ευρώπη, ιδιαίτερα με τα εθνικά μητρώα δασών, τις κυβερνήσεις, τους ιδιοκτήτες, τις Όμικρον, να αναπτύξουμε την πολιτική μας, όποια και αν είναι αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάμελ. Και εμείς θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και να τα λάβουμε υπόψη γιατί πρόκειται για μια ευρεία δημόσια διαβούλευση που θα τα λάβουμε υπόψη μας ε, πριν εκδώσουμε τη δική μας έκθεση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μάρκους Λίτνερ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Δάση, το EFI. Είναι εδώ ο κύριος Λίτνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να κάνω την παρουσίαση αυτή. Θα ξεκινήσω με θέματα που αφορούν την έρευνα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες ε, περιφέρειες της Ευρώπης. Η παρουσίαση βασίζεται στη δουλειά που κάναμε το 2008 για τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας σε μια μελέτη που αποκαλείται ε, επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος για τα ευρωπαϊκά δάση και επιλογές για την προσαρμογή. την έκθεση χρειάστηκε να την διαρθρώσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων συνθήκων που ισχύουν σε διάφορε περιοχέ τη Ευρώπη. Και όπω είπα και προηγουμένω, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των περιοχών και πρέπει να εξετάσουμε τι συγκεκριμένε επιπτώσει ε, στη βόρεια περιοχή, στην ε, ωκεάνια εύκρατη, στην υπηρετική εύκρατη και στη μεσογειακή περιοχή, όπω επίση να δούμε και τι ειδικέ λειτουργίε που ε, ισχύουν για τι ορεινέ περιοχέ. χρησιμοποιούνται πολλοί όροι και πολλές έννοιες σε βαθμό που δημιουργούν και σύγχυση. Γι' αυτό θα προσπαθήσω εδώ να σας δώσω τη γενική εικόνα, ξεκινώντας από το σημείο δεξιά, όπου αναφέρουμε τους ε, παράγοντες επιπτώσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Παραδείγματο χάρη να αυξάνεται η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακος ε, στην ε, ατμόσφαιρα. Επίσης υπάρχει άνοδος σημείωση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις ένα παράγον, καθώς και διαταραχές που οφείλονται σε βιωτικούς ή αβιωτικούς παράγοντες. Είναι διαφορετικοί λοιπόν οι παράγοντες ε, ανάλογα με την περιφέρεια και επηρεάζουν διαφορετικά τα δάση και την ευαισθησία των δασών στην κλιματική αλλαγή σε κάθε περιφέρεια. Έχουμε εδώ αυτό τον όρο λοιπόν στο κέντρο που λέει ευαισθησία κάθε περιφέρεια στους βασικούς παράγοντες που έχουν επίπτωση στα δάση οι επιστήμονες πάντοτε ε, ανησυχούν για το πόσο θα αλλάξει το κλίμα. Είναι ένας από τους ε, παράγοντες που μας ανησυχούν. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη ευαισθησία των δασών, αλλά δεν είναι μεγάλη κλιματική αλλαγή, δεν αυξηθεί δηλαδή πολύ η θερμοκρασία, μπορεί να μην έχει τόσο, σημασία, τόσο μεγάλη σημασία. Και οι δύο παράγοντες μαζί όμως θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη επίπτωση ε, και θα επηρεαστεί και η παραγωγή ξυλίας και οι άλλοι παράγοντες. Μιλάμε επίσης ε, για το ευάλωτο των δασών. Τι σημαίνει αυτό. Ε, αν τα δάση μας έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν, αν έχουν μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα, θα έχουμε ε, λιγότερο ευάλωτα δάση από ότι σε μια περίπτωση που το οικοσύστημά μας δεν θα μπορούσε να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτές είναι κάποιε βασικές έννοιες που χρησιμοποιούμε στην μελέτη μας και δεν θα σας δώσω άλλου τεχνικούς όρους για να μην σας κουράσω. Θα περάσω όμως σε μια μικρή σύνοψη αυτών που αναμένουμε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή. Από την τελευταία έκθεση αξιολόγησης τη IPCC φαίνεται ότι οι αλλαγέ ε, θα είναι περίπου δύο βαθμοί, αύξηση δύο βαθμών στο δυτικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 3 βαθμοί αύξηση στην κεντρική Ευρώπη και 4 έως πέντε βαθμοί στη βόρεια αρκτική περιοχή και σε τμήματα τη Μεσογείου. Από δύο έω πέντε βαθμοί λοιπόν θα είναι η αύξηση τη θερμοκρασία και είναι αρκετά μεγάλο γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ε, ένα βαθμό θα είναι η αύξηση σε σχέση με την μηχανική περιοχή. Φαίνεται όμω θα είναι διπλάσια ή και πενταπλάσια η αύξηση στο μέλλον. Ακόμη, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικά μοντέλα αύξηση τη θερμοκρασία. Θέρμανση το χειμώνα μπορεί να είναι μεγαλύτερη στην Ανατολική Ευρώπη, παραδείγματο χάρη, ενώ στην ε, Νότια και στη Δυτική Ευρώπη το καλοκαίρι θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση τη θερμοκρασία. Και στη Βόρεια Ευρώπη δεν, βλέπουμε, δεν αναμένουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ των εποχών του έτου. Θα υπάρχουν διαφορετικέ λοιπόν επιπτώσει στα δάση, γιατί αν είναι μεγαλύτερη ξηρασία το καλοκαίρι, θα είναι μεγαλύτερη κίνδυνη για τα δάση. Ακόμη αυξάνονται οι βροχοπτώσεις στη Βόρεια Ευρώπη, μειώνονται στη Νότια Ευρώπη σε αιτήσιο επίπεδο. Τα δάση θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις μακροπρόθεσμες αλλαγές του κλίματος και θα πρέπει να προσαρμοστούν και στο ότι αλλάζει η διακύμανση, γιατί έχουμε όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, παρατεταμένες ξηρασίες, καταιγίδε και πλημμύρες που μπορεί να είναι πιο συχνές και μπορεί να είναι και πιο έντονα φαινόμενα αναμένουμε συχνότερες ε, πλημμύρες και τέτοια φαινόμενα. Ακόμη αλλάζει η εποχιακή διαθεσιμότητα ύδατος. Αναμένουμε μεγαλύτερες βροχοπτώσεις το χειμώνα στις περισσότερες ε, περιφέρειες και μικρότερες βροχοπτώσεις το καλοκαίρι, άρα υψηλότερες ε, ξηρασίες, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για πολλά δάση. Ας περάσουμε τώρα στις ε, πιθανές επιπτώσεις που αναμένονται στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα δάση και μεγάλη διαφοροποίηση και στις επιπτώσεις επί των δασών αύξηση αναμένεται στο βορρά, περισσότερες, ε, περισσότεροι κίνδυνοι, ιδιαίτερα από πυρκαγιές στο νότο και μεγάλη κίνδυνη καταιγίδων ε, στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ευρώπης. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στα είδη των δασών και στην καταλληλότητα αναπεριφέρεια. Αυτά τα οποία τώρα λοιπόν είναι κατάλληλα μπορεί μετά από 100 χρόνια να μην συνεχίζουν να είναι εξίσου κατάλληλα για την κάθε περιφέρεια. Και 100 χρόνια είναι μια περίοδος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη διαχείριση των δασών και να προσαρμόσουμε ανάλογα τη διαχείρισή μας. Ας δούμε κάποια παραδείγματα επιπτώσεων στις διάφορες περιοχές. Στη Βόρεια Αρκτική περιοχή θα ήθελα να τονίσω ότι ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη των δασών και με τους ε, πιο ζεστούς χειμώνες ήταν, ε, υπήρχε μεγαλύτερη δυσκολία στην χρησιμοποίηση των δασών για την ε, δασοκομεία και στην χρησιμοποίηση της ξυλίας ε, λόγω των ε, εδαφών και του κατά πόσο παγώνουν τα εδάφη. Πολύ συχνά δεν μπορούν τα φορτηγά που κουβαλάνε την ξυλία να περάσουν μέσα από τα δάση. Και τέτοιες συνέπειες θα είναι ακόμη πιο σοβαρές στο μέλλον που αναμένεται ότι θα είναι πιο ζεστοί οι χειμώνες. Στην εύκρατη ωκεάνια περιοχή Υπάρχει αυξημένο κίνδυνο ε, διαταραχών από καταιγίδε και πυρκαγιέ, όπως επίσης και από την ξηρασία και γι' αυτό πάλι αλλάζει η σύνθεση των ειδών των δέντρων. Θέλουμε ήδη που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στι μελλοντικέ συνθήκες. Στην εύκρετη υπηρετική περιοχή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα με την αναδάσωση και την ε, αναγέννηση των δασών με τα υψηλότερα προβλήματα ξηρασίας το καλοκαίρι, μπορεί να έχουμε προβλήματα στα δάση τα οποία θα φυτεύουμε και υπάρχουν και προβλήματα με τέτοιες διαταραχές και σε άλλες περιοχές. Και τέλος, στην μεσογειακή περιοχή έχουμε πολλές φορές ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ σημαντικός για τη ζώνη αυτή και ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, δεν υπάρχουν ε, άλλα δάση νοτιότερα. Δηλαδή, μερικά από αυτά τα είδη δασών βρίσκονται στο όριο και αν τα είδη τα οποία τώρα υπάρχουν εκεί έχουν προβλήματα στο μέλλον, θα είναι απώλεια ως προς τη βιοπικιλότητα, διότι θα απεριμόνονται αυτές τις περιοχές και δεν θα αντικαθίστανται αυτά τα είδη δασών ε, από άλλα είδη. Ανέφερε προηγουμένω και την προσαρμοστικότητα των δασών, που είναι μια πολύπλοκη έννοια, γιατί εδώ υπάρχουν ε, δύο στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι ότι τα οικοσυστήματα αυτά καθεαυτά μπορούν να προσαρμοστούν στι αλλαγέ του περιβάλλοντο. Τα είδη των δασών λοιπόν μπορούν ε, να αλλάξουν τα ε, γενετικά τους χαρακτηριστικά από μόνα τους και προσαρμόζονται τα οικοσυστήματα, έχουν μια εγγενή προσαρμοστικότητα αλλά υπάρχουν και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες ε, που αναγκάζουν τα δάση να προσαρμοστούν. Είναι και οι δύο αυτοί παράγοντες σημαντικοί και πρέπει να τους κατανοήσουμε για να καταλάβουμε το πόσο είναι ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή τα δάση. Αυτή η προσαρμοστικότητα ποικίλει κατά πολύ αναπεριφέρεια. Στην Βόρεια Ευρώπη έχουμε εντατική διαχείριση των δασών, καινοτόμε τεχνολογίες ε, και έχουμε ε, υψηλή προσαρμοστικότητα των δασών. Στην Νότια Ευρώπη όμως οι ιδιοκτήτες των δασών και ο τομέας της οικονομίας γενικότερα είναι λιγότερο δραστήριος. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζεται η, να εφαρμόζονται μέτρα προσαρμογής ε, από πάνω προς τα κάτω ε, για να εξασφαλίσουμε τη σωστή διαχείριση και ε, επιβίωση των δασών. Εδώ θα είμαι πολύ σύντομος σε αυτή την ενότητα γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι ομιλητές που θα έχουν το ίδιο θέμα. Η προσαρμογή μπορείτε να μειώσει τις δυσμενείς επιπτώσεις ή να μας βοηθήσει ε, να βελτιώσουμε την προσαρμοστικότητα. Και αυτοί, αυτές είναι οι δύο βασικές οδοί για την μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Στη μελέτη μας εξετάσαμε επίσης και διάφορα μέτρα για την προσαρμογή των δασών. Είδαμε τι στρατηγικές υπάρχουν όσον αφορά τα δάση αυτά καθεαυτά, τη διαχείριση των δασών και την πολιτική για τα δάση. Και υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Μπορούμε ε, να πούμε ότι τα περισσότερα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να μειωθούν οι επιπτώσεις από τις διάφορες ε, διαταραχές που επέρχονται στα δάση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα που θα μας βοηθήσουν και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυξημένο κίνδυνο διαταραχών των δασών στο μέλλον. Όσον αφορά την παραγωγή ξυλίας, που επίσης ε, μας ενδιαφέρει στο θέμα της ε, προσαρμοστικότητας. Υπάρχουν μέτρα, δεν ξέρουμε όμως ποια μέτρα να εφαρμόσουμε και πότε. Ιδιαίτερα το πότε δεν γνωρίζουμε, πότε πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα είδη των δασών και πότε πρέπει να αλλάξουμε ε, κάτι στη διαχείρισή μας. Όμως ε, δεν βρήκαμε καθόλου πληροφορίες για το πώς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη διαχείρισή μας για να διασφαλίσουμε το οικοσύστημα. Δεν είμαστε ακόμη λοιπόν σωστά προετοιμασμένοι για την κλιματική αλλαγή όσον αφορά τα οικοσυστήματα. Είσαι επίμετρον λοιπόν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί μεγάλου κινδύνου, αλλά και ανοίγει και κάποιε ευκαιρίε. Η προσαρμοστικότητα είναι υψηλότερη στη βόρεια αρκτική περιοχή και στι ωκεάνιες εύκρατε ζώνε, αλλά ιδιαίτερη υποστήριξη χρειάζεται στι μεσογειακές περιοχές και στην εύκρατη υπηρετική περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Λίνερ για την ομιλία σας και σας ευχαριστώ και του δύο προλαλήσαντες γιατί ε, τηρήσατε το Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ε, πολύ σημαντική η δήλωσή σας ότι ε, ακόμη υστερούμε στην ε, χορήγηση ε, οικολογικών υπηρεσιών και τώρα το λόγο θα δώσω στον κύριο Βίνκελ που θα μας παρουσιάσει ε, το έγγραφό του ήταν η βάση για τη δουλειά της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ για την, ε, τα καλά σας λόγια. Θα μιλήσω για τις ε, επιλογές που έχει η πολιτική μας για την προστασία των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιζόμαστε σε μία μελέτη του Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ, του Ινστιτούτου για τα Δάση και το άλλο είναι το Οικολογικό Ινστιτούτο του Βερολίνου. Γενικός στόχος, στόχος των μελετών αυτών είναι να εξετάσουμε τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Κομισιόν για να για να εκπονήσει μια κοινοτική προσέγγιση για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών και για να εκτιμήσει τις δυνατότητε για μια κοινοτική πρωτοβουλία. Φυσικά δεν μπορώ να μιλήσω για όλα όσα αντιμετώπισαν αυτές οι μελέτες, άρα περιορίζουμε σε τέσσερα. Δάση και πολιτική δασών στην Ευρώπη, εισαγωγή, ε, ανάγκη για δράση σε κοινοτικό επίπεδο, επιλογές, δυνατότητες για την μελλοντική πολιτική δασικής προστασίας και συμπεράσματα. Και σε άλλες ε, εκδηλώσεις έχω κάνει αυτή την παρουσίαση, αλλά επειδή βλέπω πολλά νέα πρόσωπα μεταξύ των συμμετεχόντων, ελπίζω ότι οι περισσότεροι θα αποκομίσετε κάτι από αυτή την παρουσίαση καινούριο. Πρώτον, Το να μιλήσουμε για δάση στην Ευρώπη είναι ίδιο με το να μιλήσουμε για διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά τα δάση, την εκμετάλλευσή τους, ε, τις πρακτικές, τον τρόπο διαχείρισης ε, των δασών. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φορείς, ε, διαφορετική δομή διαχείρισης. Οπότε έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Επίσης, οι, μηχανισμοί ελέγχου και εφαρμογής ε, άλλοτε είναι περισσότερο, βασίζονται περισσότερο στην αγορά, αλλού είναι πιο βολοταριστικοί, ενώ άλλες προσεγγίσεις θέτουν προτεραιότητες σε διάφορους τομείς που θα μπορούσαμε να τους ε, περιγράψουμε ως λειτουργίες των δασών. Και τέλος, το θέμα είναι αν αντιμετωπίζουμε οικονομικά ή οικολογικά τα δάση. Που θα βασίσεις ε, την πολιτική σου, παίζει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων σου. Όμω υπάρχουν κοινέ προκλήσει παντού στην Ευρώπη. Οικολογικέ, για παράδειγμα. Κλιματική αλλαγή, μείωση τη βιοπικιλότητα, οι εκπομπέ και αποθέσει. Επίση υπάρχουν ε, κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση και την ε, ευρωπαϊκή διάσταση του κλάδου των αγορών για τα δάση. Και υπάρχει και κοινωνική αλλαγή ε, γενικότερα στην Ευρώπη. Μερικές νέες προκλήσεις, ε, μερικές νέες απαιτήσεις για τη χρήση των δασών για παράδειγμα όσον αφορά τη διασκέδαση και ψυχαγωγία, δεν είναι και τόσο καινούργιες. Όταν αναλύουμε λοιπόν την δασική πολιτική σε διάφορες χώρες, βλέπουμε δύο σαφείς διαφορετικές προοπτικές. Μία προοπτική θα μπορούσε να είναι η εμπορευματική ας πούμε, ο τομέας ε, των, ε, του κλάδου δηλαδή, των ε, επιχειρήσεων που ασχολούνται με το δάσος και η άλλη είναι η προσέγγιση της διαχείρισης που τον εκπροσωπούν, την εκπροσωπούν αυτή την προοπτική, οι μη κυβερνικέ οργανώσεις κτλ. Βέβαια δεν είναι μαύρο-άσπρο. Αλλά είναι ε, ένας διαχωρισμός που μας επιτρέπει να δούμε τις δύο πλευρές. Κυρίως εκφράζεται αυτή η διαφορά όσον αφορά την άποψη για τα δάση, πώς αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, πού υπάρχουν μεγαλύτερες ανησυχίες, ποιες είναι οι αιτίε των απειλών. Ας δούμε λοιπόν είναι εμπορευματική προσέγγιση. Εδώ το δάσος αντιμετωπίζεται ως πόρος. Οι βιομηχανίες ενδιαφέρονται φυσικά για την υγεία του δάσους, την σταθερότητα, την ζωτικότητα και ανάπτυξη και τελικά το πόσο κερδοφόρα ή μάλλον καλύτερα να καλύτερα πούμε πόσο παραγωγικά είναι τα δάση. Οπότε οτιδήποτε απειλεί την ε, παραγωγικότητα είτε είναι φυσικό ή όχι, δηλαδή αν οφείλεται και στην ανθρώπινη δραστηριότητα, λαμβάνεται υπόψη. Από την άλλη μεριά, αυτό που, εκεί που αντιμετωπίζεται ως δυνατότητα το δάσος, το δάσος αντιμετωπίζεται ως οικοσύστημα, Οπότε όλα τα ε, ζώντα όντα, ε, που αυτό που περιλαμβάνει φυσικά και τα ζώα, ε, θεωρούνται σημαντικά. Οπότε η προσέγγιση γίνεται μέσω της προσοχής στην βιοπικιλότητα, τη δυναμική της και τις απειλές. Και εδώ θεωρείται ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή οι φυσικές απειλές δεν θεωρούνται απειλές. Αυτό βέβαια έχει επιπτώσει για το πώ αντιλαμβανόμεθα την προστασία των δασών. Και για ποιο λόγο θέλει να προστατεύσει το δάσο. Και ποιου κινδύνου θέλει να αντιμετωπίσει. Και πώ. Η δασική πολιτική της Ένωσης έχει χαθεί άραγε σε αυτήν την πολυμορφία. Δεν είναι δεσμευτική η άμεση δασική πολιτική, αλλά αυτό σημαίνει πως είναι ε, αρκετά ευλίγιστη. Η έμεση πολιτική δασών μοιράζεται σε πολλούς τομείς, τον ενεργειακό τομέα, περιφερειακή ανάπτυξη, προστασία της φύσης. Υπάρχουν λοιπόν πολύ διαφορετικοί στόχοι της δασικής πολιτικής, χωρίς να έχουν σαφώς καθοριστεί προτεραιότητες. Και η εφαρμογή τους είναι πολύ άνηση, γιατί Υπάρχουν ε, κάποια νομοθετήματα, αλλά δεν είναι δεσμευτικά. Υπάρχουν βέβαια και οικονομικοί λόγοι, αλλά κυρίως είναι ότι πολλά μέτρα είναι εθελοντικά. Πρέπει λοιπόν να εκπονήσουμε μια πιο συνεκτική άποψη για την προστασία των δασών. Ας δούμε λοιπόν τα διάφορα επιχειρήματα. Για ποιους λόγους πρέπει σε επίπεδο ένωση να προστατεύσουμε τα δάση για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα για οικολογικούς λόγους, αλλά και οικονομικούς, αλλά και πολιτικούς. Η οικολογική βέβαια προσέγγιση ασχολείται με την διασυνοριακή φύση πολλών απειλών. Άρα χρειάζεται πιο συντονισμένη πολιτική σε επίπεδο ένωσης. Αλλά είναι διαφορετικά τα βιοσυστήματα των δασών από τη μία άκρη της Ευρώπης στην άλλη, άρα μάλλον ε, είναι ένα επιχείρημα κατά της εντελώ εναρμονισμένης άποψης. Από την άλλη μεριά έχουμε Ευρωπαϊκή Κοινή ε, Οικονομική Ένωση και ενιαία αγορά. Αυτοί οι, στόχοι, αυτοί, οι λόγοι είναι επιχείρημα υπέρ μια πιο εναρμονισμένης πολιτική. Αν έχει κοινή αγορά, χρειάζεται και κοινού κανόνε. Αλλά κάποιες ε, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι ο κλάδος από χώρα σε χώρα είναι πολύ διαφορετικός. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα στους κοινοτικούς στόχους και στην ε, υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την ε, απώλεια βιοπικιλότητας. Ενώ από την άλλη μεριά οι ενοποίηση σε άλλους τομείς δημιουργούν δυσχέρειες στην ενοποίηση του δασικού τομέα της αντιμετώπισης. Ενώ από την άλλη μεριά οι απαιτήσει τη κοινωνία και η αντιμετώπιση τη δασική πολιτική είναι διαφορετικέ στην Ένωση. Και κάτι που είναι μια απλή πολιτική δήλωση, αν κοιτάξουμε το παρελθόν, δεν υπάρχει αρκετή πολιτική υποστήριξη για μια πιο ενιαία πολιτική σε επίπεδο Ένωση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για δράση, αλλά η κατάσταση αποτιμάται διαφορετικά από πολλούς, γι' αυτό χρειάζονται διαφορετικές αναλλακτικές. Μία πρώτη θα ήταν να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε την παρούσα προσέγγιση. Βασισμένη στην αρχή της επικουρικότητας, απλώς να βελτιώσουμε την ε, επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δασικών πολιτικών. Δεύτερον, η επιτήρηση των ε, δασών στην Ευρώπη. Περισσότερο τονίζουμε την ε, εναρμόνιση της αντιμετώπισης για να υπάρχει περισσότερη ενότητα. Τρίτον, η προσέγγιση της οδηγίας για ε, πλαίσιο για τα δάση. Θα πω περισσότερα το, στο εγγύς μέλλον. Και τέλος, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την προστασία των δασών. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία συνενώσεις των φορέων στην Ένωση για την προστασία των δασών με μακροπρόθεσμο στόχο να βασιστούμε στις βέλτιστες πρακτικές και ε, την διαδικασία προστασίας των δασών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αυξήσουμε αυτόν τον τρόπο την ε, ενότητα της πολιτικής μας. Αυτό θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα ε, επιτόπου και βεβαίως ε, υπάρχει και το θέμα της ε, κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η πολιτική. Κύριος λόγος θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για προστασία των δασών με μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή που θα ανταποκρίνεται στις διαφορετικές φυσικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στα κράτη-μέλη. Θα ήταν ε, δεσμευτική για τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να μεταγραφεί στον, ε, στην εθνική νομοθεσία. Ο κύριος στόχος είναι να διατηρήσουμε και να αποκαταστήσουμε ένα σωστό καθεστώς, μια καλή κατάσταση όλων των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030 βάσει των κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραγόντων και να μπορούν να αντίσταται τις επιβλαβείς επιπτώσεις. Η στόχη μας είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση των δασών και τις απειλές κατά των δασών, να διασφαλίζουμε βιώσιμη διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσουμε και να ανατρέψουμε την απώλεια της βιοπικιλότητας των δασών, να βελτιώσουμε την προσαρμοστικότητα των δασών στην κλιματική αλλαγή και να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να δημιουργήσουμε τα, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πολυλειτουργική διαχείριση των δασών και τέλος να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή της κοινωνίας για θέματα που αφορούν τα δάση. Όσον αφορά τώρα τα θεσμικά όργανα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Έχουμε τα κοινά μέσα προστασίας των δασών, τα οποία ε, θα αναπτυχθούν, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προστασία των Δασών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υπηρεσιών ε, για πληρωμές στα οικοσυστήματα των δασών, το Κοινό Πλαίσιο για την Βιώσιμη Διαχείριση των Δασών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Δασών. Αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και η συνεργασία μεταξύ επίπεδου κρατών μελών και επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα κοινό κατάλογο μέτρων. Σε επίπεδο κρατών, μελών έχουμε τις εθνικές απαιτήσει, δηλαδή στρατηγικέ για τις βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση των δασών δεσμευτικά πρότυπα για τη διαχείριση των δασών, προγράμματα ε, για τα δάση, προγράμματα προσαρμογής και στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή και ε, προγραμματισμός ε, με συμμετοχή όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων δασών. Όλα αυτά θα πρέπει να διατυπωθούν σε εθνικά προγράμματα διαχείρισης των δασών και προγράμματα δράσης για τα δάση. Τέλος, κάναμε και μία εξάντε αξιολόγηση, μία εκ των προτέρων αξιολόγηση των τεσσάρων επιλογών και τα κύρια αποτελέσματα είναι ότι σαφώς υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αποδοτικότητας και του εφικτού. Όσο πιο αποτελεσματική είναι μια δράση, τόσο λιγότερο εφικτή είναι. γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, συγκρούσεις ε, με καθιερωμένα συμφέροντα στον τομέα των δασών, παραδείγματο χάρη. Ακόμη, ανάμεσα στι δύο προοπτικέ που αναφέραμε, την διαχείριση με την εμπορευματική προσέγγιση ε, και αυτά τα οποία μας είπε ο κ. Χαμέλ μετά τις διαπραγματεύσεις επί της Πρασίνου Βίβλου μπορεί να υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχουν διαφορές. Τέλος, υπάρχει συνένεση για την σημασία της βελτίωσης της πληροφόρησης για τα δάση. Και πλησιάζω στο τέλος της παρέμβασής μου. Όλες οι κοινοτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να προσπαθούν να βελτιώνουν τη συμμετοχή και τη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων για να ε, υπάρχει επαρκής ισορροπία μεταξύ όλων των απαιτήσεων και με βάση όλα αυτά υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι το πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής. Παρέχει στοιχεία και πολιτική υποστήριξη σε κοινοτικό επίπεδο και θέλουμε να έχουμε κάτι σαν οδηγία πλαίσιο για τα δάση με βάση το, τη Λευκή Βίβλο και ένα σενάριο συναπόφασης. Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό το οποίο αποκαλούμε προσέγγιση εκμάθηση της πολιτικής. Δηλαδή θα πρέπει με βάση τη διαβούλευση και τη διαδικασία συμμετοχής να προσπαθούμε να καταλήγουμε σε, στο να αλληλοδιδασκόμεθα ημένα από τους ΔΕ και να έχουμε μια ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Και το τρίτο σενάριο είναι μια προσέγγιση επιλεγμένων θεμάτων να προστατεύουμε τα δάση από τις πυρκαγιές, παραδείγματο χάρη, και να μπορούμε να ακολουθούμε για κάθε θέμα μία προσέγγιση είτε βάσει του πρώτου είτε βάσει του δευτέρου σεναρίου. Εν κατακλείδη, υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις για τις λειτουργίες των δασών, για τις απειλές για τα δάση και για την ανάγκη ε, ανάληψης δράσης. Ε, έχουμε μία ευρωπαϊκοποίηση του τομέα των δασών μέσω κοινών τάσεων και προκλήσεων στον τομέα των δασών και για τις αγορές και για τα προϊόντα που αφορούν τον κλάδο. Δεν έχουμε μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν διάφορες πολιτικές που με, μερικές φορές δεν είναι συνεπείς μεταξύ τους και χρειάζεται να σκεφτούμε τις επιλογές που έχουμε, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των δασών στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Βίνκελ, σας ευχαριστούμε πολύ ε, την αξιολόγηση των διαφόρων ε, πολιτικών λύσεων. Η συμβολή σας θα είναι πολύ σημαντική στην ε, συζήτησή μας και γενικά στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο για ερωτήσεις. Έχουμε δύο βουλευτές εδώ, μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουμε την κυρία Κορτίνες και την κυρία Σούλη. Θα ήθελα καταρχήν να τις ρωτήσω εάν έχουν ερωτήσεις προς κάποιους από τους ομιλητές του πάνελ αυτού. Η κυρία Κορτίνες. Εδώ είμαι. Από τον Νότο έρχομαι. Ε, προέρχομαι από το Βορρά, αλλά μένω στο Νότο, έχω ένα σπίτι εκεί. Έχουμε πολύ καλή διάγνωση για το βορρά, όχι όμως για τον νότο. Και δεν θα μπορέσουμε με μία πολιτική να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Λυπάμαι πολύ με αυτά που άκουσα. Ζητώ να πάμε στη βάση, να περάσουμε στη βάση. Καταρχήν, έχουμε πολύ στενό ορισμό των δασών. Τα δάση είναι δέντρα όλων των ειδών τα δέντρα και τα χαμηλά δέντρα που έχουμε στη Μεσόγειο, που διατηρούν ε, ε, το, έδαφος. Αλλά πολλά από τα χαμηλά αυτά δέντρα δεν θεωρούνται δάση. Στις περιπτώσεις όπου κάποιοι τα φροντίζουν, διατηρούνται καλά και δεν υπήρχε πολλέ πρόβλημα, ποτέ πρόβλημα, όπου υπάρχουν κάτοικοι, ε, όπου, συγγνώμη, ιδιοκτήτες, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης. Το θέμα δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι και τα δέντρα παραγωγής. Όπου υπάρχει παραγωγή είναι πιο εύκολο να διατηρηθούν. Εφόσον δηλαδή παρέχουν άμεσο όφελο στου ανθρώπου γύρω τους. Για παράδειγμα, οι βελανιδιές ε, θεωρούνται δάσος αλλά και οι αμυγδαλιέ, δεν είναι. Ο καλύτερο τρόπο διατήρηση του εδάφους ε, στην ε, Μαγιόρκα είναι οι αμυγδαλιέ. Στην Ανταλουσία είναι οι ελιέ. Είναι δέντρα. Αλλά θεωρείται γεωργία αυτό, δεν θεωρείται δασοκομεία. Υπάρχει η οικολογική τάση στην Ευρώπη και ιδεολογίε οι οποίες καταδικάζουν την γεωργία, αλλά η γεωργία βοηθάει στη διατήρηση του εδάφους. Στο μέλλον, με την οικονομική κρίση, με την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να ε, διευρύνουμε τον ορισμό των δασών, να ε, συμπεριλαμβάνει και τα, ε, και τα χαμηλά δέντρα ή χαμηλά φυτά, το θυμάρι για παράδειγμα. υπάρχουν ή, το φυτό από το οποίο βγαίνουν είναι σε, από τα οποία φτιάχνανε καλάθια και, και χαλιά το μεσαίωνα. Το σπάρτο. Είναι ε, από τους καλύτερους τρόπους ε, να ε, διατηρείται σε καλή κατάσταση το έδαφος. Υπάρχουν σχετικές έρευνες, αλλά ίσως ε, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών ε, ε, να μην φτάνουν στους ανθρώπους στα πανεπιστήμια της Βόρειας Ευρώπης, στους ανθρώπους που έχουν εξουσία, σχετικές αρμοδιότητες, αλλά που δεν τα γνωρίζονται αυτά. Και συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι θα πρέπει να γίνει η διάκριση ε, ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, όπως γίνεται και στις ε, περιφέρειες ε, όσον αφορά την βιοπικιλότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια πολιτική παντού. Συγχωρήστε με, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρώτη ιδέα λοιπόν ε, είναι να γίνει η διάκριση ανάμεσα στα δάση. Ο στόχος μπορεί να είναι ο ίδιος, αλλά τα μέσα θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική συχνά ε, μπερδεύουμε τους στόχους με τα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι διαφορετικά τα μέσα εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντική η βιοπικιλότητα όπως και το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, γνωρίζουμε ποια είναι τα είδη που θα πρέπει να φυτέψουμε. Ξέρουμε ακόμα και ποια είναι πιο καλά για τη γεωργία αλλά στο μέλλον κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή τροφίμων και ε, άλλες χρήσεις. Γίνονται παράπονα ότι η ε, Ευρώπη επιδοτεί την εκρίζωση ε, λόγω της ε, γεωργίας. Είναι σκάνδαλο το ότι η Γεωργία συγγνώμη, Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για την εκρίζωση των ε, ελιών ε, ή των κλιμάτων. Ελιές 400 ετών συχνά ε, εκριζώνονται λόγω των επιδοτήσεων στη γεωργική πολιτική. Αυτό είναι σκάνδαλο. Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη με το ένα χέρι να μιλάει για τα δάση και από την άλλη να τα εκριζώνει. Στο μεσογειακό κλίμα ένα δέντρο είναι θησαυρό. Ε, χρειάζονται ε, χρόνια να μεγαλώσει ε, και χρειαζόμαστε και την ξυλία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τη μεσογειακή πολιτική. Θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά στην Πράσινη Βίβλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχωρήστε με που παθιάζομαι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σούλη θα ήθελε να προσθέσει κάτι ώστε να απαντήσουν οι ομιλητές του πάνελ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, είσαστε τόσο αφοσιωμένοι στο θέμα ε, και μήπω θα μπορούσε η κυρία Σούλη να ε, θέσει και εκείνη την ερώτησή τη, ώστε να μπορεί το πάνελ να απαντήσει ταυτόχρονα και στι δύο ερωτήσει. Νομίζω ότι συμφωνώ με την ανάλυση της Χριστίνας στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά δάση και πολλά διαφορετικά εδάφη. Εγώ είμαι από την κεντρική Γαλλία, λίγο πιο βόρεια από την Χριστίνα και έχουμε μεγάλα δάση που είναι ιδιόκτητα δάση, τα οποία τα διατηρούν, τα συντηρούν και τα εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες τους. Ε, είναι διαφορετικό το καθεστώς από ότι όταν έχουμε πολύ μικρή ε, ε, εδάφη. Ε, υπάρχουν και δάση στα οποία, τα οποία είναι αφιερωμένα στο κυνήγι. Είναι δάση που η χρήση τους είναι να αποτελούν χώρο κυνηγιού πολύ συχνά ε, φυτεύονται κονοφόρα δέντρα ε, που είναι εντελώς διαφορετικά και αντικαθιστούν άλλα δέντρα πλατήφυλλα και ε, κάνουν το έδαφος περισσότερο όξινο τα κονοφόρα. Ένα μήνυμα προς τις δικές μας περιοχές που βρίσκονται κάπου στη μέση είναι ότι όταν κάνουμε αναδάσωση θα πρέπει να χρησιμοποιούμε είδη τα οποία να βελτιώνουν τα εδάφη, να αναπτύσσονται πιο αργά, ε, ενδεχομένως έχουν λιγότερο αποδοτική εκμετάλλευση, αλλά με αυτά τα πλατήφυλλα δέντρα ε, αναπτύσσονται παραδείγματος χάρη μανιτάρια και η καλλιέργεια μανιταριών και η συλλογή μανιταριών ε, το φθινόπωρο στη δική μου περιοχή είναι μια καταπληκτική δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι η υπευθυνότητα. Η υπευθυνότητα ανήκει και στους ιδιοκτήτες των δασών που πρέπει να φροντίζουν και το υπόστρωμα των δέντρων. Όταν έχουμε καλή συντήρηση του υποστρώματος, ε, σαφώς οι φωτιές ε, μεταδίδονται πολύ πιο αργά και γι' αυτό χρειάζεται ανάληψη της ευθύνη για να υπάρχει σωστή συντήρηση ε, του υποστρώματος. Ξέρουμε ότι το να βάλει κανείς πρόβατα κάτω από τα δάση είναι πολύ χρήσιμο γιατί καθαρίζουν ε, το έδαφος. Αυτά ήθελα να πω σαν σχόλια. Πάντως συμφωνώ με αυτά που είπε η Κριστίνα και πιστεύω ότι είναι κρίμα που αυτή τη στιγμή έχουμε ε, ελιές και μάλιστα αιωνόβιες ελιές που τις, μεταφέρουν στη Βόρεια Ευρώπη για να ομορφύνουμε τους κήπους μας γιατί πραγματικά πονάει η ψυχή μου που τις βλέπω. Είναι κρίμα για τους ελαιώνες που αποψηλώνονται στο νότο και κρίμα που φέρνουν ελιές στο βορρά για να ομορφύνουν τους κήπους χωρίς να έχουν την πραγματική χρήση τους. Είναι κρίμα αυτή η όμορφη, αυτά τα όμορφα δέντρα να μεταφέρονται στο βορρά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο για τις απαντήσεις. Ποιος θέλει να απαντήσει? very Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την ε, Κριστίνα ε, Κορτιέρες που ήταν η πρώτη που παρέμβει. Ε, έχουμε συνεργαστεί όσον αφορά το ε, ε, θα έλεγα από τότε που ήμασταν νέοι, αλλά για πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και τουλάχιστον 12 ε, χρόνια. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ σήμερα και ελπίζω να το στηρίξετε αυτό όπως μας έχετε στηρίξει και στο παρελθόν και ελπίζω επίσης να έχετε επιτυχία στην προσπάθειά σας αυτή. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα, ένα θέμα που τονίστηκε ήταν τα κλίματα και, άλλα, και, και οι ελιές. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά σημειώνω αυτό που είπατε. Το θέμα είναι η συνέπεια ανάμεσα στην πολιτική μας απέναντι στα δάση και την πολιτική μας απέναντι στη γεωργία. Και πώς μπορούμε να τις ε, συνδυάσουμε αυτές τις δύο. Θυμάμαι ότι ο λόγος για την εκκρίζωση των κλιμάτων ήταν ότι ο κόσμος δεν πίνει αρκετό κρασί. Ε, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά σημειώνω αυτό που είπατε όσον αφορά την πολλαπλή αξία των δασών. Όσον αφορά τις ελιές, ε, συμφωνώ απόλυτα με την ε, περιγραφή σας. Στην πολύ πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν για την ΚΑΠ, για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, αναφέραμε ιδιαίτερα την ε, ανάγκη για στήριξη των ε, στοιχείων της ε, φύσης υψηλής αξίας και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ελαιώνες. Θα ήθελα πολύ στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου να δω μια σύνδεση ανάμεσα στην ε, δασοκομική πολιτική μας και στην γεωργική πολιτική μας. Όσον αφορά τον Βορρά και τον Νότο, ε, πραγματικά ελπίζω αυτό να μην, ε, να μην υπάρξει πόλωση Βορρά και Νότου, διότι είναι εύκολο για αυτούς που είναι υπέρ ή κατά να στηριχθούν στη γεωγραφική βάση αντί για την επιστημονική. Τα προβλήματα των δασών στον Νότο είναι, είναι οξυμένα αλλά και στον Βορρά μπορεί να έχουμε προβλήματα με τα δάση λόγω της ε, αλλαγής του κλίματος που περιμένουμε και που βλέπουμε και λόγω της εκμετάλλευσης των δασών. Εάν ε, στερήσουμε... Εάν γίνει υπερβολική η εκμετάλλευση των δασών, μπορεί να συναντήσουμε προβλήματα και στο βορρά. Σημειώνω αυτό που είπατε για τα χαμηλά φυτά. Ε, είναι σίγουρα ένα στοιχείο που περιμένουμε να δούμε στο ψήφισμα. Όσον αφορά τα δημόσια και ιδιωτικά δάση, σίγουρα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο από τα δημόσια, ε, από τα δημόσια δάση μας. Δεν θα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των ιδιωτικών δασών με την ανακοίνωση αυτή, αλλά η ανακοίνωσή μας και το σχετικό σας ψήφισμα μπορεί να μας δείξουν τον σωστό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον τομέα των ιδιωτικών δασών. Και έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες ε, δασών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ε, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται κατά βάθο και αυτό ε, μας ε, επαναφέρει στο αρχικό μας θέμα το οποίο ανέφεραν και οι δύο βουλευτές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος τελειώνει. Ε, ε, αν θέλει ο κύριος Βίνκελ ή ο κύριος Λίντερ να απαντήσουν πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, δύο παρατηρήσεις. Η καλή διαχείριση όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα μπορεί να βοηθήσει να λυθούν κάποια από τα προβλήματα του παρελθόντος. Αυτό μπορεί να ισχύει για σήμερα, αλλά θα αλλάξει τόσο πολύ το κλίμα μας ε, τα επόμενα 50 χρόνια που οι έννοιες ε, του παρόντος και του παρελθόντος ε, δεν θα ε, μας βοηθήσουν στο μέλλον. Πράγματι είναι ε, αλήθεια ότι μπορούμε σήμερα να λύσουμε κάποια από τα ε, προβλήματα του παρελθόντος, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τη φάση αυτή, διότι στο μέλλον θα πρέπει να δούμε περισσότερο προορατικά. Όσον αφορά το θέμα της ψευδούς, του ψευδούς αισθήματος ιδιοκτησίας. Ε, ε, ε, είναι αλήθεια ότι οι ιδιοκτήτες μικρών δασών δεν έχουν κάποιες δυνατότητες. Αυτό αποτελεί πρόβλημα και στο Βορρά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλες ερωτήσεις για το τμήμα αυτό της συζήτησής μας. αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις προς όλους τους ομιλητές μας στο τέλος της συζήτησης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Jacqueline McLeod, που θα μας ε, παρουσιάσει τα ευρωπαϊκά δάση στα πλαίσια της ε, UNFCCC. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να ε, βρίσκομαι εδώ. Όπως ε, Ξέρετε, γίνονται πολλές ε, συζητήσεις και είναι πολύ απασχολημένοι, πολλοί άνθρωποι του τομέα, αλλά περισσότερο θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση η οποία στόχο έχει να σας ενημερώσουμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Έτσι μπορείτε να αποκτήσετε μια αίσθηση του τι γίνεται. Να ζητήσω συγγνώμη από κάποιους ε, συναδέρφους ε, και ε, εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, διότι θα σας παρουσιάσω εξελίξεις των τελευταίων δύο-τριών εβδομάδων. Μπορεί να μην τα γνωρίζουν αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικά στοιχεία για τις συζητήσεις σας. Να ξεκινήσω λέγοντας, όπως μας είπε και ο κύριος Λίντνερ, Χάρηκα πολύ ότι χρησιμοποιείται ο τρόπος ταξινόμησης, αλλά αυτό είναι ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ε, στην Ευρώπη δηλαδή έχετε πολύ περισσότερες ε, διαβαθμίσεις ε, στην ταξινόμηση. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουμε στο παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα θέλω να καλύψω το τι κάνουν τα κράτη-μέλη όταν ξεφεύγουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και συμμετέχουν σε άλλα φόρουμ. Ε, ένα από αυτά είναι το GEO, ε, η ε, Global Environment Observations, όπου συμμετέχουν και άνθρωποι από τον διαστημικό τομέα για να, γίνουν, για να γίνει, μπορεί να γίνει παρακολούθηση της κατάστασης. Πριν τρει εβδομάδε στο Πεκίνο, στην ε, Διεθνή Υπουργική Διάσκεψη, συζητήθηκε το εξής. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει μέσω των ε, θεσμικών φορέων. Δεν ισχύουν λοιπόν οι ρυθμίσεις που ισχύουν εδώ στο Συμβούλιο, για παράδειγμα. Ήταν όμω ενθαρρυντικό το ότι πολλά κράτη-μέλη συμμετέχουν ως κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει λοιπόν συντονισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές θέσεις. Ε, και πολύ σημαντικό είναι αυτό που γίνεται σχετικά με το land cover, σχετικά με την κάλυψη της γης. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορα, διάφορα λόγκο στη σελίδα αυτή. Ε, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, υπάρχει το δικό μας ε, λογότυπο. Ε, βλέπετε το κοινό κέντρο ερευνών. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία του χάρτη αυτή, αυτού. Έχουμε τώρα κανονισμό σχετικό που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου του φετινού έτους. Όσον αφορά τα δάση λοιπόν, Υπάρχει μια σειρά θεμάτων σε διεθνές επίπεδο ε, σχετικά με το πώς ταξινομούνται τα δάση. Ένας από τους βασικούς ε, μίσο που προσπαθήσαμε να ε, ασκήσουμε την επιρροή μας είναι η ισορροπία ανάμεσα στην Ήπεθρο, την, ε, τις περιφέρειες, τους βιοτόπους, ε, τα είδη δασών κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς και βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα. Στην GEO προσπαθούμε να εναρμονίσουμε και να απλοποιήσουμε τουλάχιστον από ευρωπαϊκής πλευράς το τι θα θέλαμε να δούμε σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την πληροφόρηση. Ιδιαίτερα με τις χώρες του ΕΟΧ ε, που συμπεριλαμβάνει και την, ε, την ΕΖΕΣ, ε, την Τουρκία, τη Γρυλανδία κλπ. Μέσω της Forest Europe ή άλλων φορέων μπορούμε να φροντίσουμε να χρησιμοποιείται μια μεθοδολογία που να αναγνωρίζεται διεθνώς και που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, για τις ε, σημαντικές ε, συμβάσεις όπως είναι η UNFCCC. Βλέπετε εδώ λοιπόν έναν χάρτη που δείχνει πώς μπορούμε να δούμε τι κάλυψη δασών υπάρχει. Αυτό χρησιμοποιείται και από την Eurostat. Ένα τέτοιο χάρτη όμω δεν μα λέει πολλά. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. Επανέρχομαι όμω στην συζήτηση σχετικά με τον Νότο. Βλέπετε ότι γύρω από τη Μεσόγειο υπάρχουν πολλά δάση. Το θέμα είναι πόσο κατακαιρματίζονται τα δάση και με την εξηρασία που επικρατεί πολλά από τα δάση αυτά κινδυνεύουν. Σε επίπεδο GEO έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο που πραγματοποιείται εδώ και αρκετό καιρό που έχει να κάνει με το Forest Carbon Tracking. Τα στοιχεία αυτά εισραίουν στις εκθέσεις που δημοσιεύονται από την UNFCCC και το Red Plus. Στην υπουργική διάσκεψη σίγουρα οι εργασίες της ομάδας κρούσης αυτής αναγνωρίστηκαν ε, πολύ καλά, αλλά ε, επιπλέον παρατηρήθηκε ότι κάτι πιο σημαντικό είναι η παρακολούθηση και πληροφόρηση σχετικά με τα δάση. Εδώ συμμετέχουμε και εμείς και το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Θέλουμε να ε, παράγουμε στοιχεία τα οποία να εισβαίνουν στο RED και στο RED+. Ως άμεση χρήστες λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε οι προσπάθειες και η χρηματοδότηση που ε, εισβέει στα διαστημικά προγράμματα να χρησιμοποιείται. Και θεωρούμε ότι ο ρόλος μας είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την δημιουργία μεγάλου όγκου πληροφοριών, είτε μιλάμε για παρακολούθηση, παρακολούθηση παιδιάσμα κτλ, που να είναι άχρηστα ουσιαστικά, που να μην είναι κατάλληλα για την δουλειά που τα θέλουμε. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στα ε, παγκόσμια ή στα διεθνή αυτά προγράμματα και να δούμε πού έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες συμφωνίες, πού μπορούμε να ε, συμβάλλουμε μεθοδολογικά, πού μπορούμε να έχουμε σημαντικό διάλογο με τις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος Silver ή με άλλους ή με άλλες χώρες. Ε, προσπαθούμε λοιπόν ε, να ασκήσουμε επιρροή στα παγκόσμια προγράμματα, στα διεθνή προγράμματα. Είναι όμως πρόκληση όλα αυτά. Αποφασίσαμε λοιπόν με την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών μας, ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά προβλήματά μας. Έχουμε τους συναδέλφους μας στη Ρωσία, από την άλλη μεριά των συνόρων, ε, σε μια εποχή όπου ο διάλογος ε, είχε αποδυναμωθεί, αποφασίσαμε να αναζωογονήσουμε το διαλογο ε, Ευρώπη Ρωσία. Ήταν δύσκολο, αλλά νομίζω ότι πάλι βρισκόμαστε σε ένα ε, προορατικό επίπεδο ε, και η δασοκομεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο των διαλόγων και εντός της Ρωσίας γίνεται αναδιοργάνωση στους, σχετικού στους σχετικούς τομείς. Πριν κάποιες εβδομάδες από την πλευρά της Ρωσίας ε, η Περιβαλλοντική φορείς μετεωρολογικοί και το Υπουργείο Οικονομικών ε, ήρθαν στην Κοπεχάγη και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για τα δάση αυτά. Μιλάμε για ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών και από το διάστημα και κάποια άλλα ε, στοιχεία παρακολούθησης για να δούμε πώς θα μπορέσουμε γρήγορα να καταλήξουμε σε έναν αλγόριθμο, σε μια μεθοδολογία ε, για να μιλάμε για τις αλλαγές εντός των δασών. Αυτή είναι η πρόκληση. Δεν μιλάμε για την παραγωγή ενός χάρτη. Θέλουμε ε, να έχουμε ε, ευέλικτη χαρτογράφηση. Και παρόλα, παρότι μας λέει η διαστημική υπηρεσία, δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν μόνο από το διάστημα. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που έχουμε ένα διετές ε, πρόγραμμα εργασίας, ε, στο οποίο συμμετέχουν ε, εδώ και πρόσφατα ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ε, αρχικές επιχειρήσεις ε, είχαμε το πλεονέκτημα να συνεργαζόμαστε με διαφόρους από την ΚΑΦ και από τον ε, βιομηχανικό τομέα όσον αφορά την παρακολούθηση της γης. Τα δάση αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ. Στις συνομιλίες μας με τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται πολύ για το πρόγραμμα αυτό, στόχος μας είναι να έχουμε χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης, μιλάμε για ανάλυση 15-20 μέτρων. Στις αρχικές αυτές επιχειρήσεις ε, θέλουμε να έχουμε πραγματικές υπηρεσίες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία, από τον βιομηχανικό τομέα και από άλλους φορείς. Το Forest Layer λοιπόν είναι ένας ε, τομέας προτεραιότητας για μας. Όπως βλέπετε έχουμε τρεις ε, Βασικέ περιοχέ όπου θα γίνουν οι δοκιμές και όταν μιλάμε για δοκιμές μιλάμε ε, για ανθρώπου που θα πηγαίνουν στα δάση, να παρακολουθούν και θα βλέπουν τι θα γίνεται. Η Σουηδία λοιπόν ε, είναι ε, η μία περιοχή, έχουμε όμω και συναδέλφους από τη Ρωσία και από την Βόρεια Αμερική, από τον Καναδά. Στόχος εδώ είναι να συνδυάσουμε τις διαστημικές, τη διαστημική παρακολούθηση με την επίγεια παρακολούθηση και με τις πραγματικές συνθήκες. Ε, συγκεντρωνόμαστε στο περίοδο διότι ε, η περισσότερη δουλειά που γίνεται έχει γίνει στα τροπικά ε, δάση και όχι στα βόρεια. Άλλο πρόγραμμα που έχουν παρουσιάσει οι Ρώσοι είναι ο συνδυασμός της χαρτογράφησης με εικόνες από ραντάρ και ιδιαίτερα είναι διατεθειμένοι να ανταλλάσσουν τα μετεωρολογικά στοιχεία που έχουν από ραντάρ με μας. Και αναφερθήκατε στον ε, καιρό στη μετεωρολογία και αυτή η υψηλή ανάλυση είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την, ε, τις πυρκαγιές στα δάση και άλλα πράγματα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορέσουν να επηρεάσουν κάποια από τα θέματα που έχουμε ε, όσον αφορά την εναρμόνιση, την πληροφόρηση κλπ. Όλα αυτά ε, τα στοιχεία θα εισρεύσουν στο, στο σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών της GEO. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το βιομηχανικό τομέα, διότι η Σουηδία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία και άλλες χώρες προσυπέγραψαν ε, αυτό και ε, συμφώνησαν να υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών με ε, τις με την κατάλληλη κατανομή. Κάτι λοιπόν που παλιά ε, θεωρεί το επιστευτικό μπορεί τώρα να είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Ε, θα το αφήσω αυτό όμως στα κράτη-μέλη, πάντως θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι μερικές φορές τα κράτη κάνουν κάτι ε, σε διεθνές επίπεδο και κάτι άλλο σε ευρωπαϊκό. Δεν θα αναφερθώ υπερβολικά σε αυτό. Η βασική ιδέα είναι πάντως να μην βασιζόμαστε αποκλειστικά στα στοιχεία από το διάστημα. Έχουμε τα στοιχεία in situ, τα οποία συνδέονται με αυτές τις ε, αρχικές επιχειρήσεις ε, επίγειας παρακολούθησης. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τη χρηματοδότηση για να προωθήσουμε εντός του βιομηχανικού τομέα ε, τους εταίρους μας που θα μας παρέχουν υπηρεσίες. Αρκετοί από αυτού συμμετέχουν ήδη όσον αφορά τη χαρτογράφηση και την χρήση της γης και Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι εντός δύο ετών μέχρι το 2013 θα έχουμε τη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης ε, ως υπηρεσία σε ε, συνεργασία με μια σειρά ε, βιομηχανικών εμπορικών εταίρων και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα θέλουν τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της UNFCCC και η Ιαπωνία κάνει κάτι παρόμοιο. Στόχος είναι όταν ε, τεθούν στο ε, τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, αυτά τα διάφορα συστήματα να ε, γνωρίζουμε για τι πράγμα μιλάμε. Γνωρίζουμε ήδη ότι το σύστημα των Ιαπωνέζων δεν είναι πολύ ακριβές, ιδιαίτερα όχι όταν έχει κανείς να κάνει με τα είδη των δασών που έχουμε στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι Λοιπόν, να μην αναφερόμαστε μόνο στο περιβαλλοντικό κεκτημένο, αλλά να λέμε κιόλας ότι έχουμε ε, πολύ διαφορετικά είδη δασών στην Ευρώπη και να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Θα πρέπει να Συνεχίζουμε λοιπόν την παρακολούθηση. Πάρα πολύ σημαντικό όμω είναι και το θέμα τη ποιότητα του εδάφου. Ε, το λέμε αυτό και στην έκθεση την οποία ε, δημοσιεύσαμε χθε. Πολύ ευχαρίστω ε, θα σας απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν. Ε, πάντως ε, η ουσία είναι ότι ήθελα να το αναφέρω αυτό εδώ σε εσά ε, για να γνωρίζετε τι κάνουμε σε διεθνές επίπεδο, πέρα από αυτά που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ζακλίν, ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικά τα εργαλεία που διαθέτουμε και τα δυνητικά μας εργαλεία για τη δημιουργία πολιτικής και θα είναι σημαντικό βήμα για το μέλλον. Και τώρα θέλω να ζητήσω από τον κύριο Μπερνάρντ Γκάλεμπερ να λάβει το λόγο. Είναι υπεύθυνο και διευθύντη για τον τομέα των δασών στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Βιομηχανιών Χάρτου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Όταν κανείς ε, μιλά σε μια συνεδρίαση μετά από άλλους ομιλητές, υπάρχει ο φόβος ότι θα επαναλάβει τα ίδια πράγματα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω μια νέα προοπτική. Θα ξεκινήσω δηλώνοντας κάτι που ίσως για πολλούς φαίνεται προφανές. Ε, είναι κάτι το οποίο αναφέρεται από τους επιστήμονες στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης ε, του IPCC, της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και τα βασικά σημεία ήταν ότι είναι σημαντική η βιώσιμη διαχείριση των δασών που πρέπει να συμβάλλει στο μετριασμό και την αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα ε, παράγοντας ε, βιώσιμη ετήσια παραγωγή ξυλίας, ινών και ενέργειας από τα δάση. Αυτό είναι αυτό που τελικά θα δώσει το υψηλότερο βιώσιμο όφελος όσον αφορά το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για να τα επιτύχουμε αυτά χρειάζονται δάση τα οποία θα είναι σωστά διατηρημένα και εδώ έχουμε μια σημαντική πρόκληση. Συνοψίζοντας αυτή τη διαφάνεια θα ήθελα να πω Συνήθως λέμε ότι τα δάση μας δίνουν τέσσερα ωφέλη, που τα λέμε τα τέσσερα S από τις τέσσερις λέξεις στα αγγλικά που αρχίζουν από S. Αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακος στα δάση, αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακος σε προϊόντα ξύλου, αποθήκευση υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από βιομάζα και υποκατάσταση των μη ανανεώσιμων πρώτων υλών με ξύλο. Και σαφώς η προϋπόθεση είναι η αηφόρος διαχείριση των δασών. Γνωρίζουμε ότι τα δάση υπόκεινται σε διάφορες απειλές. Απειλές όπως τις έχουμε εντοπίσει είναι τα διάφορα παράσιτα και ασθένειες και αυτό το ξέρουμε από τα δάση στο Δυτικό Καναδά που έχουν ε, πληγεί από παράσιτα φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, καταιγίδε, ξηρασίες, ε, παγετός, κατολιστήσεις. Αστάθεια των δασών, διότι το έδαφος γίνεται περισσότερο ασταθές λόγω της θέρμανσης. Και πιο μακροπρόθεσμα ενδέχεται να αλλάξει το μείγμα των ειδών ή να αλλάξει η τοποθεσία των ε, δασών, και από μια μελέτη που έχει γίνει στη Γερμανία έχουμε πάρει αυτό το slide και νομίζω ότι αφορά τα δάση οξιάς στη Βαβαρία για το που βρίσκονται σήμερα και το που θα βρεθούν με την αλλαγή του κλίματος. Όλες αυτές οι απειλές σαφώς έχουν επιπτώσεις επί των δασών. Και εδώ έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Αλλάζουν τα δάση, έχουν επίπτωση στην αλλαγή του κλίματος, η αλλαγή του κλίματος έχει περαιτέρω επιπτώσει στα δάση. Αλλάζει η αλληλεπίδραση δασών και υδάτινων πόρων. Η βιοπικιλότητα επίσης επηρεάζεται και έχει επιπτώσεις επί των δασών όσον αφορά ε, το νεκρό ξύλο, την πανίδα, τους οικοτόπους. Τα δάση συμβάλλουν στο μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, αλλά σιγά σιγά θα έχουν μικρότερη επίπτωση σε αυτό τον τομέα. Ενδέχεται να αυξηθεί η δέσμευση άνθρακα από τα δάση. Θα είναι περισσότερο ευάλωτα τα δάση από κινδύνους ε, θανάτου των δασών και από την καταπώνηση των δασών. και ενδέχεται να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα των δασών. Αυτό που σημαίνουν όλα αυτά είναι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε την διαχείριση των δασών. η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να είναι προσαρμοσμένη στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα είδη που επιλέγονται και φυτεύονται πρέπει να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική λογική παραγωγή βιομάζας και ανέφερε ο κύριος Χάμελ ότι η βιομάζα πρέπει να επιτύχει το στόχο του 20% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τα δάση πληρούν διάφορες λειτουργίες που αφορούν τη βιοπικιλότητα, την αναψυχή, την προστασία των υδάτινων πόρων. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την ανάγκη για φόρο διαχείριση των δανών των δασών, συγγνώμη. Και όπως είπε και ο κύριος Λίντνερ, πρέπει να προσαρμόσουμε την διαχείρισή μας πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα δοθούν από τις κατάλληλες πολιτικές που θα χρησιμοποιούν. Προς το παρόν υπάρχουν πολλά τα οποία διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Προσπάθησα να δω την νομοθεσία που ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη και είδα ότι χρησιμοποιούμε διαφορετικού όρου. Πολλέ φορέ χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέσα μέτρηση. Οι μονάδε μέτρηση δεν είναι ίδιε. Και πραγματικά η Κομισιόν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αν μπορούσε να ενοποιήσει αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη για τη διαχείριση των δασών. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε επικαιροποιημένα δεδομένα και ο τρόπος με τον οποίο τηρούνται τα εθνικά αρχεία δεν είναι ενοποιημένος. Επίσης υπάρχει κατακαιρματισμός αρμοδίων φορέων. Σε άλλα κράτη είναι αποκεντρωμένη η διαχείριση, σε άλλα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Δεν είναι καθόλου σαφές ποιος κάνει τι σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Και έχουμε και πάρα πολλές μη συντονισμένες πολιτικές για πολλούς άλλους τομείς εκτός από τα δάση που έχουν επιπτώσεις επί των δασών. Στη διαφάνεια αυτή προσπάθησα να αναφέρω ορισμένα, όχι όλα, ορισμένα από τα μέσα πολιτικής που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα από αυτά δεσμευτικά, αλλά όχι, και προσπάθησα να τα συνδέσω με την αρμόδια γενική διεύθυνση ή με τον αρμόδιο οργανισμό. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον 7 διαφορετικές γενικές διευθύνσεις αναφέρονται εδώ και θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τον κατάλογο αν θέλαμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι σαφώς υπάρχει ανάγκη συντονισμού και αν δεν γίνεται αυτός ο απαραίτητος συντονισμός, το αποτέλεσμα θα είναι ότι μπορεί παράλληλα να αυξάνεται η αγρανάπαυση και η κινητοποίηση της βιομάζας για να επιτύχουμε του στόχους του 20% για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Τι θα κάνουμε με τις πρώτες ύλες. Θα χρησιμοποιούμε αυστηρά κριτήρια αηφόρου ανάπτυξης ενώ παράλληλα δεν θα έχουμε δεσμευτικά εναρμονισμένα κριτήρια για τη βιομάζα. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, μπορούμε να επηρεάσουμε μόνο την δέσμευση του άνθρακα και όχι την υποκατάσταση ενεργειακών πόρων και στην πρόσφατη ανακοίνωση για την κοινή γεωργική πολιτική η λέξη δάσος αναφέρεται μόνο μία φορά, ενώ τα δάση καλύπτουν το 40% των εδαφών της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης. Δείτε το και μόνοι σας στο διαδίκτυο. Έψαξα εγώ στην κοινή γεωργική πολιτική και η λέξη δάσος αναφέρεται μία φορά. Σαφώς λοιπόν κάτι λείπει. Τα δάση συνεισφέρουν σε τόσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο μία φορά αναφέρονται στο κείμενο της ανακοίνωσης. Τι πολιτικές χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε καλύτερες γνώσεις, καλύτερα δεδομένα, καλύτερα στατιστικά στοιχεία και ανάλυση αυτών και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ακόμη χρειάζεται εξισορρόπηση των λειτουργιών των δασών. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις σίγουρα θα χαμογελάσουν ακούγοντάς το, γιατί χρόνια τώρα το συζητούν. Χρειάζεται ισορροπία στις διάφορες λειτουργίες των δασών, ούτως ώστε να έχουμε αηφόρο διαχείριση των δασών. Ακόμη πρέπει να ενισχύσουμε τα ωφέλη και τις υπηρεσίες ε, των δασών και να χρησιμοποιούμε ε, τα δάση και την ξυλία καταρχήν για την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και να τα καίμε μόνο όταν δεν έχουμε άλλη πιο επικοδομητική χρήση. Ακόμη πρέπει να διασφαλίσουμε το συντονισμό και την συνεκτικότητα των δεδομένων. Ανέφερε και ο κύριος Βίνκελ ένα σενάριο με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και παράλληλα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Να ορίσουμε ποιο κάνει τι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να μην ξέρουμε ποιο είναι υπεύθυνο. Κάποιο λοιπόν πρέπει να είναι αρμόδιο, τουλάχιστον ξέρουμε σε ποιον να στείλουμε τα παράπονά μα. Και παράλληλα να μην ξαναρχίσουμε από την αρχή, να μην προσπαθήσουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά για την προώθηση της αηφόρου διαχείρισης των δασών και είναι κρίμα να μην τα λάβουμε υπόψη αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην ΣΕΠΗ, στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των βιομηχανιών ε, χάρτου υπάρχουν, ε, ε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και συνεχίζονται οι συζητήσεις αυτές και έχουν οριστεί διάφορα σημασιολογικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Τι σημαίνει αηφόρος, τι σημαίνει συντονισμός, τι σημαίνει πολιτική, τι σημαίνει πλαίσιο, ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Και έχουμε παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν ισχύει μόνο στην Ευρώπη, αλλά ισχύει και σε εθνικό και ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο, ότι τα περισσότερα όργανα που είναι αρμόδια για το δάσος και τη δασοκομεία έχουν την αρμοδιότητα, αλλά πολλές φορές δεν έχουν την εξουσία να υλοποιήσουν την πολιτική για την οποία έχουν αρμοδιότητα. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε, πάντοτε είναι πιο εύκολο να πούμε τι δεν θέλουμε παρά τι θέλουμε. Αυτό που δεν θέλουμε λοιπόν είναι ένα τεράστιο μηχανισμό όπως η κοινή γεωργική πολιτική, αυτό που είχε κάνει η κοινή γεωργική πολιτική για τα δάση. Θέλουμε μια πολιτική κοινού πλαισίου, αλλά όχι ένα βαρύ μηχανισμό. Στην χαρτοβιομηχανία βρισκόμαστε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση, γιατί η βιομηχανία μας είναι παγκόσμια, πρέπει να ανταγωνιστούμε με τη Βραζιλία, με την Κίνα και παράλληλα αναζητούμε πόρους ε, δίπλα μας, σε μικρά δάση που είναι μικρές ιδιοκτησίες, πολύ κοντά στις ε, χαρτοβιομηχανίες μας. Βρισκόμαστε λοιπόν κάπου ανάμεσα στα δύο. Έχουμε παγκόσμιες προκλήσεις από τη μια πλευρά και από την άλλη τους πόρους μας που αναζητούμε ε, στη γειτονιά μας. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να αποφύγουμε τις αντιφάσεις στην πολιτική μας. Αυτά τα οποία ήδη γίνονται και γίνονται σωστά δεν πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να μην υπάρχει επικάλυψη. Να δούμε τι κάνει Forest Europe και να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση των δασών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μπερνάντο Καλαμπάρ. Ήταν πολύ σαφές αυτό που είπε για τον κατακαιρματισμό των υπάρχουσων πολιτικών ε, για τα δάση και την ανάγκη συντονισμού. Δεν θέλει κοινή γεωργική πολιτική. Ανέφερε και την ε, προσέγγιση πλαισίου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βέρλεντος. που εκπροσωπεί την Φέρν και την Life θα μας μιλήσει για τον ρόλο της βιοπικιλότητας ε, στην ενίσχυση της ε, αντοχής των δασών ε, στην αλλαγή του κλίματος. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ την Φέρν και την Μπέτλα εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδέρφους μου, ε, και Παρή, που με βοήθησαν να ετοιμάσω την σημερινή παρουσίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και μια σειρά μη κυβερνητικών οργανώσεων που μας παρήχαν τις ε, εικόνες για την ε, παρουσίαση αυτή για να σας δείξουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Πρόκειται για μη από την ε, Ουγγαρία, Γερμανία, Σουηδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Όλοι θα γνωρίζετε ότι η BirdLife είναι πολύ μεγάλη οργάνωση με πολλούς εταίρους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δάση ελπίδας που ε, στόχο έχει να ε, που ε, υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων για δάση στις τροπικές περιοχές αλλά συνεργάζεται και με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ευρώπης για θέματα πολιτικής δασών. Η ΦΕΡΝ είναι πολύ μικρή μη κυβερνητική οργάνωση και ε, εργάζεται υπέρ των καλών πρακτικών δασοκομεία και ε, συντηρήσεων των δασών στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας αναφέρω διάφορα θέματα σήμερα. Καταρχήν ε, να σας μιλήσω για την βιοπικιλότητα και την αλλαγή του κλίματος. Κατόπιν πολύ σύντομα να αναφερθώ στην πολιτική δασών της Ευρώπης. Μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τις πυρκαγιές, ε, την ε, διαχείριση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια σύντομη ανάλυση της ε, πράσινης βιβλίου για την προστασία των δασών και κατόπιν να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Δεν ξέρω εάν ήδη είχατε το χρόνο να κοιτάξετε την ανάλυση της διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους για την Πράσινη Βίβλο. Κυρίως βασίζεται σε μη κυβερνικές οργανώσεις, υπάρχουν όμως και ε, ε, απαντήσεις από ε, πολίτες, ιδιώτες και ζητείτε εδώ διατήρηση της βιοπικιλότητας. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω κάποια από τα κείμενα που εμφανίζονται στην έκθεση αυτή που ετοιμάστηκε για το CBD και που έχει να κάνει με την αντοχή των δασών και την βιοπικιλότητα. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι όταν ε, μιλάμε για βιοπικιλότητα, μιλάμε για βιοπικιλότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για ε, επίπεδο οικοσυστημάτων, μιλάμε και σε επίπεδο ειδών ε, ή, ακόμα και γενετικού υλικού. Γενικά τα τα τεχνητά δάση είναι πιο ανθεκτικά, γι' αυτό κατά τη γνώμη μας ε, οι πολιτικές ε, και τα μέτρα ε, που που συντηρούν τα φυσικά δάση έχουν πολλά ωφέλη. Επίσης, ε, οι φυτίες ε, και τα τροποποιημένα φυσικά δάση θα αντιμετωπίσουν ε, μεγαλύτερους κινδύνους απολειών μεγάλης κλίμακας από την αλλαγή του κλίματος. Η έκθεση επίσης αναφέρει έναν κατάλογο μέτρων μετρίασης των κινδύνων δεν θα σας διαβάσω τον κατάλογο αυτόν, αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω ότι επικεντρώνονται οι παρατηρήσεις στη διατήρηση της γενετικής επικιλότητας και την διεύρυνση ήδη υπαρχουσών δικτύων την διαχείριση δασών με οικολογικό τρόπο, την ε, μείωση του φυσικού ανταγωνισμού με τον έλεγχο των ε, επεκτατικών ειδών, ε, να μειώσει την χρήση των μη τοπικών ειδών και την αύξηση της βιοποικιλότητας. Δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση. Ο κύριος Βίνκελ έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση και όπως και ο Μπερνάρντ Ντε Κολομπέρ θα ήθελα απλά να τονίσω ότι και εμείς θεωρούμε την ε, δασική πολιτική ένα πολύ μπερδεμένο δίκτυο. Υπάρχουν πολλές πολιτικές που επηρεάζουν τα δάση και βλέπουμε ότι η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο αφήνει το πεδίο ανοιχτό για ε, ασυνέπεια. Βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε, στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τα δάση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχο έχει να δώσει εξίσου ίσο βάρος σε εμπορικές ε, και περιβαλλοντικές ε, σε εμπορικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα, αλλά δεν τα, δεν καταφέρνει. Υπάρχει κενό ανάμεσα στην διαχείριση των δασών επί χάρτου και του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Στην πράσινη βίβλο είχαμε και κάποια νούμερα, τα οποία βλέπετε εδώ στην οθόνη, για να σας δείξω ότι τα δάση της Ευρώπης ε, χάνουν υγεία και βιοπικιλότητα. Έχει υπονομευτεί η δυνατότητα των ε, δασών όσον αφορά την αντίσταση στην ε, αλλαγή του κλίματος. Οι πολιτικές έχουν μειώσει την δυνατότητα των δασών να ε, αντίστανται στην, στην αλλαγή του κλίματος υπό το φως των εξελίξεων είναι πολύ σημαντικό για μας να εκπονήσουμε ένα αποτελεσματικό, εμπεριστητωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την ε, προστασία των δασών. Χωρίς ε, τον απαραίτητο συντονισμό θα συνεχίσουν να διαβρώνονται τα δάση καθώς και η δυνατότητά τους ε, να να μετριάσουν την αλλαγή του κλίματος και να μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε σε αυτήν. Ε, ο Μπόρις και η Πάρη... Okay, και ο Πάρης με βοήθησαν πολύ ε, για το ε, επόμενο κομμάτι της παρουσίασής μου. Η πράσινη βίβλος καταλήγει ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ των συμμετεχόντων ότι τα δάση της Μεσογείου θα επηρεαστούν περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος. Η Life ε, δημοσίευσε φέτος μία έκθεση που λέγεται Against the Green, η οποία υπάρχει και στην ε, ιστοσελίδα τους, η οποία επικεντρώθηκε σε δύο βασικά θέματα. Η αποτελεσματική διαχείριση των δασών ε, τελικά αποτελεί κενά λόγια, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Στο δεύτερο μέρος της έκθεσής τους παρουσιάζουν κάποιες περιπτώσεις πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα οικοσυστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις περιπτώσεις επικεντρώνεται σε μια περιοχή Natura 2000 στην Περοπόννησο, στην Νότια Ελλάδα, που επλήγει από μια τεράστια πυρκαγιά το 2007. Συνήθως η διαχείριση μετά από μια πυρκαγιά ε, συμπεριλαμβάνει πολύ ακριβές παρεμβάσεις όπως είναι η ε, η απομάκρυνση των ε, νεκρών ε, δέντρων και την ε, επαναφύτευση. Αυτό όμως δεν επιτρέπει στα δάση να αποκατασταθούν με φυσικό τρόπο. Με απλά μέτρα χαμηλού κόστους και με πληροφοριακή εκστρατεία έχουμε μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο να βοηθήσουμε να αποκατασταθούν τα δάση μετά από μια πυρκαγιά. Οι επαναλημμένες πυρκαγιές σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελέσουν σημαντική απειλή ε, για μια περιοχή, αλλά το να βελτιώσουμε την αποκατάσταση μετά τις πυρκαγιές ε, είναι εξίσου σημαντικό με την, ε, με την αποτελεσματική διαχείριση για την αποφυγή των πυρκαγιών θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην προώθηση της ε, κατάλληλης χρήσης της γης, ώστε η ε, τόποι αυτή να μην είναι ευάλωτη στις πυρκαγιές. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Θα σας δείξω κάποιες εικόνες διαφόρων ε, καταστάσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σας δείξουν την έλλειψη συνέπειας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση. Επίσης θα σας δείξει το χάσμα ανάμεσα στην ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών στο χαρτί και στην πράξη. Πιστεύουμε ότι η πολιτική δεν συμβάλλει ούτε στην ε, βιοποικιλότητα, ούτε ε, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κλίματος. Όπως είπε ήδη η κυρία Μακλέιτ, η ΕΕ παρουσίασε χθε μια αξιολόγηση του περιβάλλοντος της Ευρώπης. Ε, όσον αφορά τα δάση, ε, κατέληξε η μελέτη ότι ε, τα περισσότερα δάση της Ευρώπης αποτελούν αντικείμενο πολύ σημαντικής εκμετάλλευσης. Μόνο το μισό περίπου, λιγότερο από το μισό θεωρείται ότι δεν έχει πειραχτεί από ανθρώπους βλέπουμε κατακαιρματισμό των ε, υπολείπων δασών, ε, κάτι που, ε, κάτι που εξηγεί εν μέρη στην, κατάσταση, στην κακή κατάσταση των δασών. Βλέπετε εδώ μια δορυφορική εικόνα από την κεντρική Σουηδία, στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν δάση, δυστυχώς όμως στην εικόνα αυτή. Ίσως δεν είναι πολύ σαφές αν κάθεστε πίσω. Φαίνεται όμως ότι, ε, ότι δημιουργούνται ότι χρησιμοποιούνται για ξυλία όλο και περισσότερα ε, μέρη των ε, δασών αυτών. Η Πράσινη Βίβλος δείχνει ότι τα περισσότερα δάση στην Ευρώπη έχουν την ίδια ηλικία. Τα περισσότερα είναι μεταξύ 60 ε, και 80 ετών. Βλέπετε εδώ το, την ηλικία των δασών στην Σουηδία, όπως επίσημα έχουν ε, παρουσιαστεί από τις Σουηδικές Αρχές. Ε, βλέπετε λοιπόν στον άξονα Χ τα δάση, τις κατηγορίες ηλικιών, συγγνώμη, και στον άξονα Ψ βλέπετε τον αριθμό των εκταρίων. Αν κοιτάξετε καλά ε, το διάγραμμα αυτό θα δείτε ότι στην αρχή οι κατηγορίες ηλικιών ε, καλύπτουν ε, δεκαετίες, ενώ προς το τέλος 40 χρόνια. Μια μη κυβερνητική οργάνωση στην Σουηδία άλλαξε κάπως την διαφάνεια αυτή και έτσι αλλάζει η συνολική εικόνα. Ουσιαστικά πολύ λίγες περιοχές έχουν μείνει όπου τα δάση είναι απείραχτα. Όσον αφορά την ε, συμβολή στην επίτευξη των στόχων βιοπικιλότητας ε, και αλλαγής του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την αποκατάσταση των δασών, τη δάσωση. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα της Ουγγαρίας όπου χρησιμοποιήθηκαν χρήματα για την δάσωση από το 2007 μέχρι το 2009. Ε, χρησιμοποιήθηκε όμως κυρίως για μη εγγενή είδη και βλέπετε εδώ πέρα ε, ένα είδος ιδιαίτερα επεκτατικό, το ρομπίνια. Ε, το οποίο ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, καθιστά πολύ δύσκολη την, την αποκατάσταση των δασών. Πρόκειται για την γαζία. Επίσης, η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επηρεάζει πολύ τα δάση, θα προωθήσει πολύ την παραγωγή ε, βιοενέργειας ε, και αναμένεται να διπλασιαστεί η χρήση βιομάζας, κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα τα δάση εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να τονίσω δύο θέματα. Στο μεταξύ όμως υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν τι κενό υπάρχει ανάμεσα στην προσφορά και στην ζήτηση όσον αφορά τις μελλοντικέ ανάγκες ε, στον ε, τομέα παραγωγής ξυλίας ε, και βιομάζας. Θα υπάρχει λοιπόν σημαντικό κενό. Δεν... Θα υπάρχει αρκετή ξυλία και για τους δύο τομείς, το παραγωγής ξυλίας δηλαδή και βιομάζας. Φοβούμαστε ότι θα δούμε εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων υλοτομία. Και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ε, σωστή διαχείριση των δασών. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, ανθεκτικότητα των δασών ε, στην αλλαγή του περιβάλλοντος. Βλέπετε εδώ μια εικόνα από ε, την Σουηδία. όπου αφαιρείται και το τελευταίο κομμάτι του κορμού του δέντρου για να χρησιμοποιηθεί για βιομάζα. Ε, αυτό ε, επηρεάζει και το περιβάλλον και το, την ποιότητα του εδάφους. Πηδάω κάποια παραδείγματα και φτάνω στην Πράσινη Βίβλο. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι ε, επικροτούμε την Πράσινη Βίβλο σε μεγάλο βαθμό, διότι επικεντρώνεται στα δάση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε ότι τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να συγκεντρώσουν την προσοχή μας. Υπάρχουν κάποια πολύ ισχυρά σημεία στο έγγραφο αυτό. Πιστεύουμε ότι δίνει μια πολύ καλή επισκόπηση ε, των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος στα δάση αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Επίσης αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στη γνώση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με δεδομένα που έχουν να κάνουν με τα δάση. Κάποια αδύναμα σημεία είναι ότι επικεντρώνεται πολύ στην αλλαγή του κλίματος κάτι θετικό. Ελπίζαμε όμως να δούμε περισσότερες ε, διασυνδέσεις ανάμεσα στην αλλαγή του κλίματος ε, και την βιοπικιλότητα. Θα μπορούσε επίσης ε, να αναφέρει το έγγραφο περισσότερο τις ασυνέπειες όσον αφορά την πολιτική. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν η Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών ε, άρχισε να ετοιμάζεται. Λίγες μέρες πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέδωσε την ε, έκθεση για τη βιομάζα που συνδέεται με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μπορούσε να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στις δασοκομείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολυλειτουργικότητα και βιώσιμη διαχείριση των δασών. Το έγγραφο δεν ε, αναγνωρίζει ότι έχουν αποτύχει οι έννοιες αυτές και ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση και ότι μάλιστα ε, δεν υπάρχει αρκετή ανάλυση των συνεπειών των πρακτικών δασοκομείας ε, τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά για παράδειγμα την βιοπικιλότητα, την ε, δέσμευση του ε, διοξιδίου του άνθρακα και πολλά άλλα θέματα. Να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Κάτι ξέχασα, έπρεπε να ε, βιαστούμε κατά την ετοιμασία της παρουσίας αυτής. Φυσικά χαιρόμαστε που το, που η Πράσινη Βίβλος ε, έχει να κάνει με το σύστημα πληροφόρησης ε, για τα δάση και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να διασφαλίσουμε την ύπαρξη σωστών συστημάτων πληροφόρησης. Εάν θέλουμε να αναλάβουμε δράση σε κάποιους τομείς, κάτι τέτοιο είναι απόλυτα απαραίτητο και στον τομέα της βιοπικιλότητας. Όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από το απλά να βελτιώσουμε τα συστήματα πληροφόρηση για τα δάση πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο ώστε να διασφαλίσουμε την ε, αυξημένη προστασία των δασών και πιστεύουμε ότι οι ε, συζητήσεις που θα γίνουν στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σημαντικό κενό ανάμεσα στο τι έχουμε επί και στο τι γίνεται επί Ζητάμε από τους διάφορους φορείς, τους ιδιοκτήτες των δασών, ε, την, ε, το σχετικό βιομηχανικό τομέα και τις αρχές να έχουν μια σχετική συζήτηση, δηλαδή το τι γίνεται στην πράξη στη διαχείριση των δασών. Ε, η σωστή διατήρηση των δασών θα βοηθήσει στο μετριασμό των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, τις, ε, θα βοηθήσουν και στην διατήρηση της βιοπικιλότητας ε, και χρειάζεται να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της ε, παρούσας πολιτικής για τα δάση. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν οι πολιτικές αυτές να είναι πιο συνεκτικές και πώς μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των δασών. Πιστεύουμε επίσης ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να αναλυθεί ώστε να εντοπιστούν ε, ελλείψεις ε, στην χρηματοδοτική δομή ε, και για να βελτιωθεί η χρηματοδότηση. Εάν τα δάση ε, πρέπει, αν τα, δάση της Ευρώπης θέλουμε να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος και να μετριάσουν την αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε και εσάς και το φορέα που εκπροσωπείτε, τη Fern και την Life. Ε, δύο μη κυβερνητικέ οργανώσεις παρουσιάστηκαν με την ε, παρουσίαση αυτή και είναι πολύ καλό το ότι συνεργάζονται αυτές οι οργανώσεις. Σημειώσαμε τα μηνύματα που ακούσαμε για τις δυσκολίες, ε, για την ε, αποτελεσματικότητα, για, τη χρήση, ε, για την απαραίτητη χρηματοδότηση, για την προστασία των δασών. Και ελπίζω ότι θα γίνουν και πράξη αυτά τα οποία ξέρουμε ότι υπάρχουν θεωρητικά. Μετά από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη συζήτηση. Ε, θα έχουμε διερμηνία μέχρι τις 4.30. Αν χρειαστεί να συνεχίσουμε μετά τις 4.30 θα πρέπει να συνεχίσουμε μόνο στα αγγλικά χωρίς διερμηνία. Θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Μάτα να λάβει το λόγο για την πρώτη ερώτηση. Και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Κρήτον. Έφτασα καθυστερημένη και δυστυχώς ε, δεν άκουσα όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που ήδη συζητήσατε. Ως ε, Ευρωβουλευτής από τη Σουηδία, γιατί είδαμε και κάποιες φωτογραφίες από τη Σουηδία, το λέω αυτό. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν καταρχήν διαφορές μεταξύ των 27 κρατών μελών. Στην ε, Σουηδία το 75% του εδάφους καλύπτεται από δάση. Και έχουμε πολλά καλά παραδείγματα για τη διαχείριση των δασών και στη Σουηδία και σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα και είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε την βιοπικιλότητα και πού πρέπει να μπουν οι διαχωριστικές γραμμές. Ακούσαμε παραδείγματα, αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε και άλλα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Υπάρχουν χώρες και περιοχές κυρίως που ζουν από την δασοκομεία. Ζουν από τα δάση και γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξουμε και να μην καταστρέφουμε τα δάση μας. σε 50 ή 100 χρόνια δεν θα έχουμε πόρους αν καταστρέφουμε τα δάση. Είναι όπως και η αλία που πρέπει να προσέξουμε στην εκμετάλλευση των δασών. Ίσως όμως επαναλαμβάνω πράγματα που ήδη είπατε κατά τη συζήτηση στην οποία δεν ήμουν παρούσα. Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε πού βάζουμε τη διαχωριστική γραμμή. Και το λέω αυτό ζώντας σε μια περιοχή της Ευρώπης ε, που, ε, όπου τα δάση έχουν οικονομική σημασία και έχουν σημασία για την απασχόληση και με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το περιβάλλον. We, Όντως έγινε μια μεγάλη συζήτηση για διάφορα θέματα και έγινε η παρουσίαση δύο εκθέσεων από την EFI, από το Ινστιτούτο για τα Δάση και από το Ινστιτούτο του Φράιμπουργκ, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν για τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Και θα ήθελα τώρα ε, να ακούσω από τους συμμετέχοντες είτε σε αυτό το πάνελ είτε στο προηγούμενο, αν θέλετε να απαντήσετε στις ανησυχίες που εξέφρασε η συνάδελφος. Ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές.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 δεν θα απαντήσω ακριβώς για το θέμα των διαχωριστικών γραμμών, γιατί δεν είμαι εγώ ειδικό για να σα πω πού πρέπει να βάλουμε τη διαχωριστική γραμμή. Θα επαναλάβω όμως την ανησυχία του κλάδου, γιατί σας είπα ότι θέλουμε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών. Η βιομηχανία την οποία εγώ εκπροσωπώ έχει αναλάβει δεσμεύσεις πολλές φορές για την αηφόρο διαχείριση και εκμετάλλευση των πρώτων υλών. Και σαφώς το γνωρίζετε αυτό από τη Σουηδία, διότι ανακυκλώνουμε περισσότερο. Οι πόροι τους οποίους χρησιμοποιούμε δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ακριβώς διότι χρησιμοποιούμε περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά και πιστοποιημένα υλικά. Η πιστοποίηση είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι είμαστε μια υπεύθυνη βιομηχανία και όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε. Θέλω να τονίσω την ανησυχία μου για το ότι υπάρχουν εξελίξεις σε πολιτικές σε άλλους τομείς που δεν ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Και επανέρχομαι στο θέμα της βιοενέργειας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Και δεν υπάρχουν κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα. Υπάρχει ένας κλάδος που κάνει ό,τι μπορεί για να είναι όλο και περισσότερο υπεύθυνος και να τηρεί τις αρχές της αηφόρου διαχείρισης και από την άλλη πλευρά δεν ζητείται η ίδια υπευθυνότητα στον ενεργειακό τομέα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια τέτοια ανανεώσιμη ενέργεια δεν είναι αναγκαστικά πράσινη, αν δεν υπάρχουν διασφαλίσεις που απαιτούνται. Δεν ε, είναι κόκκινη γραμμή, διαχωριστική γραμμή, αλλά είναι ένα κόκκινο φως προειδοποίησης αυτό που λέω. Θα ήθελα να ακούσουμε περισσότερες ερωτήσεις να ακούσουμε λοιπόν περισσότερες ερωτήσεις, ε, αν δεν έχετε αντίρρηση, και κατόπιν οι ομιλητές θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, διότι πραγματικά τελειώνει ο χρόνος μας. Παρακαλώ, όποιο παίρνει το λόγο, αν μπορείτε να πείτε το όνομά σας και ποιον φορέα εκπροσωπείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγομαι Νέλα Μίκολα από την Κόπα Κοσέκα και χαίρομαι που με προσκαλέσατε στην εκδήλωση αυτή. Εκπροσωπώ ε, γεωργούς και ιδιοκτήτες ε, ιδιοκτήτες δασών. Ίσως θα μπορούσα να σας δώσω την ε, προοπτική των ιδιοκτητών των δασών. Πιστεύουμε ότι τα δάση είναι σημαντικός φυσικός πόρος και υπάρχουν πολλές πτυχές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ε, κοιτάμε το δάσος ε, στο σύνολό του. Υπάρχουν πολλές πτυχές, ε, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Σε σχέση με άλλους φυσικούς πόρους, τα δάση είναι ένας πόρος που είναι γενικά στη διάθεσή μας. Να μην ξεχνάμε και την πτυχή της απασχόλησης. Υπάρχουν ε, δάση που εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους. Η ε, διαχείριση των δασών λοιπόν έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε τα θετικά αποτελέσματα στην βιοπικιλότητα αλλά και όσον αφορά την ε, ανθεκτικότητα σε φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πυρκαγιές. Η ε, ενεργός διαχείριση των δασών ε, έχει να παίξει ρόλο στην πρόληψη τέτοιων γεγονότων. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους άλλους φυσικούς πόρους. Έχουμε τα δάση ως συμβολή στην ε, αλλαγή του κλίματος ε, διότι δεσμεύουν ε, το διοξίδιο του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και την υλοτομία ως δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα. Οποιοδήποτε μέσο λοιπόν αναπτυχθεί το οποίο να επηρεάζει τα δάση θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συντονισμού και εξέτασης του ε, τομέα των ε, δασών στο σύνολό του. Εάν δεν είναι ανταγωνιστική ε, η υλοτομία δεν θα μπορεί να παρέχει και τα πλεονεκτήματα που μπορεί. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ομιλία του κυρίου Γκαλομπέρ. Η Forest Europe υπάρχει, είναι μια πρωτοβουλία. Πώς θα ληφθεί αυτή η υπόψη από την Κομισιόν κατά τον καθορισμό των μελλοντικών εργασιών. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στην μελλοντική κυνηγεωργική πολιτική και πώς αναγνωρίζει τη συμβολή των δασών. Ε, για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Στην ανακοίνωση Είδαμε ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται μία φορά η λέξη δάση. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε να λαμβάνονται υπόψη στην ε, πολιτική αυτή στο μέλλον. Αλλά πιο σημαντικό είναι να προωθηθεί η χρήση του ξύλου. Είναι ένας πόρος φυσικός πόρος με θετικές συνέπειες στην αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να δούμε τις θετικές συνέπειες της χρήσης της ξυλίας και πώς λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν το θέμα αυτό σε σχέση με τους άλλους φυσικούς πόρους που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Μάρτιν Κερλίχη από την Ελλάδα. Εκπροσωπώ την Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. ή δύο σχόλια. Καταρχήν, τα ξένα επιθετικά είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αποτελούν ένα κίνδυνο προς τα ευρωπαϊκά δάση και χαιρετίζω αυτό που ανέφερε ήδη η κυρία Τόση στην παρέμβαση της. Υπάρχουν στοιχεία ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει θετικά ε, την ε, εισαγωγή ορισμένων ε, ειδών όπως τα ελάνθους στα δάση της Βορείου Μεσογείου καθώς και σε κάποια δάση της Νοτιού Μεσογείου. Υπάρχουν δηλαδή ήδη κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τρόπο επίλυσης αυτών των προβλημάτων που οξύνονται. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα ε, να θίξω αφορά την ε, προστασία των ε, δασών. Το πρώτο θέμα αφορούσε τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Το δεύτερο αφορά την προστασία από τις πυρκαγιές. Στο πέρασμα των χιλιετηρίδων, μετά την νεολιθική εποχή ιδίω, οι πυρκαγιές των δασών επηρεάζουν τα δάση αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο που είναι τμήμα της οικολογικής διαδοχής ε, οικοτόπων. Δεν εννοώ με αυτό ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε τα δάση από τις πυρκαγιές. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πρέπει το γεγονός αυτό να το συμπεριλάβουμε στον προγραμματισμό της προστασίας των δασών. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύουμε τα δάση από την πυρκαγιά έχοντας κατά νου αυτούς τους, αυτές τις οικολογικές παραμέτρους, να μην τις αγνοούμε. Το ότι οι πυρκαγιές των δασών μερικές φορές Ε, αργούν να ε, συμβούν στα δάση μπορεί να δημιουργήσει ε, πρόβλημα ω προ την ένταση των πυρκαγιών. Να είναι πολύ μεγάλε, πολύ έντονε, και να δημιουργήσουν ακόμη και απώλεια ανθρώπινων ζώων. Ε, ορισμένα ε, δάση όπως ε, ένα είδος πέθκης είναι προσαρμοσμένο στην τακτική εναλλαγή πυρκαγιών γιατί στην περιοχή της Μεσογείου οι πυρκαγιές παρουσιάζουν ένα φαινόμενο εναλλαγής και η προστασία των δασών μερικές φορές επηρεάζεται θετικά από εναλλασσόμενες πυρκαγιές. Ευχαριστώ. Οι επόμενοι ομιλητέ παρακαλώ να είναι πολύ σύντομοι για να έχουμε χρόνο και για τι απαντήσει και να έχουμε και πιο πολλέ ερωτήσει. Ο κύριο Σκούλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια μικρή ερώτηση, μάλλον περισσότερο δήλωση είναι. Παρακαλώ πείτε μας ε, ποιον εκπροσωπείτε. Εκπροσωπώ το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ε, Ευρωπαϊκής Μεσογειακής ε, ε, περιβαλλοντικής υπηρεσίας και εκπροσωπώ γενικά έναν φορέα που εκπροσωπεί πολλές μεσογειακές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μου είπαν, αλλά δεν είχα το χρόνο το ελέγξω, ότι τα βελγικά δάση είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του βασιλέα Λεοπόλδου σε εποχή κρίσης που ήταν τόσο σημαντική η ανεργία που ο μόνος στόχος ήταν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ίσως να έχουν έτσι τα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να το ελέγξουμε. Ξεκινώ με αυτό διότι πιστεύω ότι Η διαχείριση που χρειάζεται για τα δάση θα βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον για τουλάχιστον κάποιους από αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι τον Απρίλιο του 1987 οργανώσαμε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τότε Βελγικής Προεδρίας την πρώτη διεθνή, το πρώτο διεθνές συμπόσιο για τη διαμόρφωση μιας κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής για πρόληψη και ε, αντιμετώπιση των ε, πυρκαγιών των δασών στην ε, Μεσόγειο. Το 1987 ήταν αυτό και τότε Ακόμα και με την όξινη βροχή, που αποτελούσε ακόμα πρόβλημα τότε για τα βόρεια δάση, Και όπως είπε ο κ. Χάμελ, ελπίζω να είμαστε πιο σοφοί τώρα πια, να μην βλέπουμε ε, τα πράγματα ως αποτέλεσμα πώλησης, ε, πόλωσης βορρά και νότου. Το πρώτο που είχαμε, το μόνο που έχουμε από τότε είναι η ευρωπαϊκή δάση δεδομένων για τις πυρκαγιές που υπάρχει ακόμα. Αυτό είναι θετικό. Αλλά ε, φτάνω τώρα στο έγγραφο και το θέμα των ε, τριών επιλογών. Προφανώς από τα όσα είπα πιστεύω σε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, διότι μια τέτοια θα έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από μειονεκτήματα. Και πιστεύω ότι οι λόγοι γι' αυτό είναι καταρχήν ότι τα δάση αποτελούν διαπραγματευτικό σημείο για την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, καταπολέμηση της ε, αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει να έχουμε κοινή φωνή. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα σχετικά με την εξή διάκριση. Μιλάμε για την προσαρμογή, αλλά θα πρέπει να δούμε τα δάση ως μέσο προσαρμογής. Άλλο θέμα είναι η προσαρμογή των δασών. Μιλάμε εδώ για δύο ξεχωριστά θέματα και τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, το πιο σημαντικό για τον Βορρά και τον Νότο είναι το θέμα του νερού. Και όσον αφορά τη διασφάλιση του νερού και όσον αφορά την ε, πρόληψη των πλημμύρων, ε, υπάρχουν τα δάση τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν μιλάμε λοιπόν για την προσαρμογή των δασών στην αλλαγή του κλίματος, μιλάμε για τα δάση που είναι απαραίτητα για τη δική μας προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την αντιμετώπιση του θέματος του νερού. Γι' αυτό θα πρέπει το θέμα αυτό να ε, συνδεθεί στενά και με το έγγραφο ε, για την προσαρμογή Το άλλο θέμα είναι τα μικρά δάση. Τόσα θέματα αναφέρατε. Ναι, είναι σημαντικό να έχουμε τους ελαιώνες. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στους ελαιώνες ηλικίας εκατοντάδων ετών και αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα σήμερα, τις... την φύτευση των νέων ελαιώνων. Θα πρέπει να γίνει εδώ διάκριση. Θα σταματήσω. Άλλα 30 θέματα είχα να αναφέρω, αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ε, δούμε και γραπτώς αυτά τα σχόλια για να ληφθούν υπόψη οι αρκούντος. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εκπροσωπώ το γυμνάσιο τη Αντορίνη. Δεν υπάρχει μετάφραση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο στα αγγλικά. Πέρασε, είναι και μισή. Μισή μεταφραστέ. Θα σου επειδή υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί θα μπορούσαν να μείνουν μεταφραστέ για αυτή την ερώτηση για μόνο. Ε... Νομίζω ότι μπορείτε να προχωρήσετε αυτή την ερώτηση μόνο. Εντάξει. Θα το πούμε στα ελληνικά. Μπορεί να γίνει και μετάφραση από εδώ, από τη συνάδελφο. Α. Λοιπόν, ε, θα είμαι πολύ σύντομο. Οι κλιματικέ αλλαγέ επηρεάζουν ε, σίγουρα και θα επηρεάσουν. οι μεταφραστέ λένε μόνο την ερώτηση. Θα, γιατί πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ναι. τη δουλειά του. Πολύ σύντομο λοιπόν. Ε, και επηρεάζουν και θα επηρεάσουν ε, τα δάση μας οι κλιματικές αλλαγές. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής για ένα φαινόμενο μάλλον ελληνικό για τις πυρκαγιές που έχουν στόχο την ε, οικοπεδοποίηση και τι προβλέπετε για τις ε, αναδασώσει, για γιατί σίγουρα προστασία του δάσους θα είναι αν ε, υπάρχει υποχρέωση της αναδάσωσης. Και μια και μίλησε η κυρία Κορτίνες για τα χαμηλά φυτά, θα εκφράσω μια απορία. Ε, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδότησε κάποια στιγμή την εκρίζωση των αμπελώνων και μάλιστα θεωρώ το αρχαιότερο αμπελώνα του κόσμου που είναι της Σαντορίνης και ένα φαινόμενο που δυσαρέστησε πάρα πολλούς ε, Σαντορινιούς και εμάς φυσικά και το σχολείο και τους μαθητές μας. Βέβαια ο μόνος ε, λόγος που βλέπουμε ήταν ότι οι ανταγωνιστές μας δεν μπορούσαν να συναγωνιστούν το υπέροχο κρασί μας και βρήκαν έναν τρόπο να καταστρέψουν τον αμπελώνα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. There was someone else asking for the floor. Yes. Hello, my name is Satu Antianen and I work for the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 So it makes me sad if you say something like this. Thank you very much. I will take a question from Michael Stramopoulos, another MEP, if he wants to take the floor. Μιλάμε αγγλικά μόνον. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω περισσότεροι είναι Έλληνες. Δεν έχω κάτι να προσθέσω